Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας με το σημείο 21, Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό έτος 2003. Στις 4 Απριλίου δημοσιεύθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού και θα γίνει η παρουσίαση τον Ιούλιο μάλλον η γνωμοδότηση. Θα γίνει τώρα η πρώτη ανταλλαγή απόψε. Επί της γνωμοδοτήσεως Ριβελίνη. Έχετε το λόγο κύριε Σιγητά για να μας παρουσιάσετε τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. E- Σας ευχαριστώ και να απευθείας στο θέμα. Ο προϋπολογισμός για το 2013 από την Σκοπιά μου ως απαιτεί να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις. Γι' αυτό θελήσαμε να κάνουμε κάποιες ε, προτάσεις για τις πιστώσεις που προβλέπονται για το κεφάλαιο Αλία και σε κάποιες δημοσιονομικές γραμμές. Σε πρώτη ανάγνωση, η ελάχιστη αύξηση του προπολογισμού στο σύνολό του, στο 2% δηλαδή, δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί για να καλύψει τις δημοσιονομικές ανάγκες όλων των κλάδων. Άρα, ένα τέτοιο ε, κλάδο, όπω ε, αυτό τη Αλία που είναι στρατηγική και πρωταρχική σημασία, τελικά ε, πλήττεται. Συγκεκριμένα, <clears throat> στο πλαίσιο του δημοσιονομικού προγράμματο για το 2013 δεν ε, προβλέπονται, δεν δεσμεύονται επαρκεί πιστώσει για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και για το υποστηρικτικό τη πρόγραμμα. Δεν θα αναπτυχθούν περαιτέρω. Η δημοσιονομική γραμμή 11 σημείο ουσιαστικά δεσμεύει ε, πιστώσεις πληρωμών για το 2013 που δεν είναι αρκετές. Ζητώ λοιπόν να μάθω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Όσο το δυνατόν συντομότερα. Ε, για ποιο λόγο προβλέφθηκε αυτό το ποσό και ελπίζω όσο το δυνατόν συντομότερα να ανακτήσουμε για αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα μία ε, συγκεκριμένη πίστοση. Η ίδια μέρημνα αφορά την ε, κοινή αλληλευτική πολιτική. Συγκεκριμένα, τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασχοληθεί με την συντήρηση και την αξιοποίηση του αλλιευτικού υδρολογικού τομέα την, της γραμμής 1107 στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και του δυσχερούς ε, Διαστήματο που διανύουμε θα πρέπει να στηριχθεί. Ένα άλλο σημείο που πλήττεται είναι αυτό της ε, αγοράς της αλίας με τη γραμμή 11.0,2 και με μείωση 20% σε σχέση με το 2012. Έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες που είχαν καθοριστεί για την περίοδο 2007-2013 και στο πλαίσιο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, μεταξύ άλλων η στήριξη των επιχειρησιακών δομών, η ανάπτυξη επιχειρήσεων που είναι οικονομικά εύρωστες, όλες αυτές οι προτεραιότητες δεν μπορεί να μας οδηγούν σε μια τέτοια μείωση. Θα προκληθούν τεράστιες ζημιές σε αυτόν τον σημαντικότατο κλάδο. Σημειώνω επίσης με ικανοποίηση τις αυξήσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας, για τους στόχους σύγκλησης γραμμή 110612 και τη μή σύγκλησης, σημείο γραμμή μάλλον 110613. Εκεί προβλέπεται αύξηση 33.600.000 ε, ευρώ περίπου για τους στόχους σύγκλησης και 11.200.000 ευρώ για τους στόχους εκτός σύγκλησης. Σημειώνω επίσης τη σημασία που αποδίδεται στο ταμείο, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλία και την προσαρμογή των ε, κοινοτήτων ε, ψαράδων που δεν, για μη βιομηχανικούς σκοπούς, οικολογικότερες μορφές παραγωγής και βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον, ευθύ αμέσω θα πρέπει να προβλεφθεί στον προϋπολογισμό το, η συνολική πρικοδότηση ε, ταμείο Ταμείου για την Αλία, στη γραμμή 1106, λαμβάνοντα υπόψη και την προσχώρηση τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Ούτω ώστε να μην τύχουν δυσμενού μεταχειρήσει ούτε τα κράτη-μέλη που ήδη ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε να μειωθούν οι εκταμιεύσει του, ακριβώ επειδή θα προσχωρήσει και η Κροατία αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, θα ήθελα να μάθω γιατί ε, αποφασίστηκε τεράστια περικοπή, περίπου 15% για την διακυβέρνηση, την governance των κοινών ε, αγορών της Αλίας, γραμμή 11.0,4. Θα πρέπει να, συντηρηθούν, να διατηρηθούν μάλλον τουλάχιστον στο επίπεδο του 2012 οι πιστώσεις για την συντήρηση και την αξιοποίηση των αλληλευτικών πόρων στη γραμμή 1107. Οι περικοπές που προβλέπονται για τον προπολογισμό του 2013 επηρεάζουν σημαντικούς ε, τομείς της αλίας και δεν θα επιτρέψουν τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτού του τόσο σημαντικού κλάδου. Ακριβώς την περίοδο της ε, οικονομικής κρίσης που διανύει η Ευρώπη. Για αυτούς τους λόγους και αναμένοντας ε, αιτιολογημένες ε, απαντήσεις για αυτές τις σημαντικότατες περικοπές, είναι σημαντικό να επανεξετάσουμε όλες τις δεσμεύσεις και τις πιστώσεις ε, που έχουν να κάνουν με το κεφάλαιο 11. Ευχαριστώ πρώτη. πρέπει να τα του συναδέλφου. Ευχαριστούμε κύριε Ριβελίνη. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους όμως, να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ίσως έπρεπε να είναι και η πρώτη. Εν πάση περιπτώσει, ας ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σα παρουσιάσω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2013. Να ξεκινήσω με κάποιες γενικές παρατηρήσεις ως προς το πλαίσιο και μετά να επικεντρωθώ σε ορισμένα στοιχεία της πρότασης για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλία και θα προσπαθήσω τέλος να απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις του κ. Ριβελίνη. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πριν από ένα μήνα περίπου το σχέδιο προπολογισμού τη και ο Επίτροπο Λεβαντόφσκι ήρθε αμέσω στην Επιτροπή Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρουσιάσει αυτό το σχέδιο. Όπω είπε ο κ. Ριβελίνη, Όντως περίοδους, διανύουμε περίοδους κρίσης και η πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2003 έγινε με οδηγούς δύο βασικές ιδέες. Καταρχήν, την ιδέα του ρεαλισμού, την αρχή του ρεαλισμού, ώστε οι βασικές πληρωμές για το 2013 έλαβαν υπόψη την προηγούμενη εφαρμογή των πιστώσεων Άλλη κατευθυντήρια αρχή του προπολογισμού είναι η ευθύνη, η υπευθυνότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Γιατί οι αναλήψεις υποχρεώσεων αποτελούν νομικές βάσεις για μελλοντικές πληρωμές. Οι σημερινές αναλήψεις υποχρεώσεων, οι σημερινές υποσχέσεις είναι αυριανές πληρωμές και γι' αυτό ε, αποφασίσαμε για το 2013 αναλήψεις υποχρεώσεων ε, να παραμείνουν σταθερές και άρα, όπως είπε ο κύριος Ριβελίνη, η αύξηση στις δεσμεύσεις υποχρεώσεων ε, περιορίζεται στο 2%, στον τιμάριθμο δηλαδή, στο ποσοστό του πληθωρισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει πάνω από 150 δις ε, για αναλήψη υποχρεώσεων και 138 περίπου δισεκατομμύρια για πληρωμές. Το σχέδιο προϋπολογισμού δεν καλύπτει το κόστος της προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό το κόστος ήδη έχει συζητηθεί και αποτελεί τμήμα του δημοσιονομικού πακέτου που συμφωνήθηκε στην διάσκεψη της ένταξης. Εμείς θα υποβάλουμε ένα διορθωτικό για την προσχώρηση της Κροατίας κατά τις αρχές του 2003. Εγκαίρως πάντως, πριν την ένταξη, τότε θα υποβληθεί ο διορθωτικός προϋπολογισμός και μάλιστα εμπρόθεσμα, γιατί όπως ξέρετε η ένταξη της Κροατίας προβλέπεται για τον Ιούλιο του 2013. Τώρα επανέρχομαι στους συγκεκριμένους τίτλους και δημοσιονομικές γραμμές. Τα προτινόμενα ποσά για τις θελάσσιες υποθέσεις και την αλία αντιστοιχούν σε ένα σταθερό πλαίσιο για τα προγράμματα και τις δράσεις του τίτλου αυτού. Το συνολικό ποσό των ε, αναλήψεων υποχρεώσεων είναι πάνω από ένα δις και των πληρωμών 835 εκατομμύρια για το 2013. Περιλαμβάνονται εδώ οι διοικητικές δαπάνες, δαπάνες διαχείρισης και προσωπικού δηλαδή. Τα ποσά είναι σχετικά σταθερά, αν τα συγκρίνουμε με το 2012. Υπάρχει μια μικρή μείωση κατά 1,4% σε αναλήψεις υποχρεώσεων που εξηγείται όμως από την κατάσταση στη θαλάσσια πολιτική. Και υπάρχει και αύξηση κατά 3,6% στις πιστώσεις πληρωμών. Τώρα, αν δούμε τις δαπάνες και την κατανομή τους στις διάφορες πολιτικές, βλέπουμε ότι τη μερίδα του Λέοντος την έχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελίας. Εκεί οι δεσμεύσεις είναι τα 2 τρίτα του προϋπολογισμού. Εδώ διαπιστώνουμε μια αύξηση σε σχέση με το 2012, όπως ε, παρατηρήσε και ο κύριος Ριβελίνη, μια αύξηση 2,3%. Έχουμε δηλαδή 686 εκατομμύρια ευρώ τώρα για το 2013. Επίσης, οι πιστώσεις πληρωμών και αυτές αυξήθηκαν αισθητά, αν τις συγκρίνουμε ε, με το 2013 βλέπουμε αύξηση 7,3% για το ΕΤΑ σε σχέση με το 2012. Και το θέμα των επαρκών απιστώσεων πληρωμών είναι ένα ζήτημα που επισήμανε η Επιτροπή σας Πολάκης και το λάβαμε υπόψη. Αυτή η αύξηση στις πληρωμές θα καλύψει και τις ενδιάμενες πληρωμές που θα γίνουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελίας και που θα μπουν στην κανονική τους πορεία το 2013. Το πιο σημαντικό τμήμα του προπολογισμού αφορά τη διεθνή διάσταση των δραστηριοτήτων μα Εκεί η αναλήψη υποχρεώσεων για τις διεθνείς αλληλευτικές συμφωνίες και το δίκαιο τη Θάλασσα είναι 14% του συνολικού προϋπολογισμού. Ε, αυτό θα, το ποσό θα καλύψει και τα ποσά των αλληλευτικών συμφωνιών, των FPA, αλλά και τα κονδύλια που θα διατεθούν για τα πρωτόκολλα Τώρα, τα ποσά που ζητήσαμε για το αποθεματικό μας αντανακλούν τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διασφαλίσουμε ε, σταθερές αλληλευτικέ δυνατότητες σε πολλές αλληλευτικέ συμφωνίες για το 2013. Τώρα, για αυτό το διεθνέ κεφάλαιο έχουμε ε, πιστώσεις για ε, υποχρεωτικές και προαιρετικές συμμετοχές σε FMO και σε οργανισμούς του ΟΗΕ και φυσικά βελτιωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση και βιώσιμη ε, διαχείριση της αλίας, διαχείριση της αλίας σε διεθνές επίπεδο. Τώρα αναφερθώ σε δύο σημαντικά τμήματα της αλληλευτικής μας πολιτικής. Τη συντήρηση και τον έλεγχο. Αυτά είναι κεφάλαια παρόμοια σε σημασία Έχουμε εκεί κάποιες ε, μικρές μειώσεις στις πιστώσεις πληρωμών και θα σας εξηγήσω γιατί. Σε ό,τι φορά τη συντήρηση υπάρχει μια μικρή μείωση, 4% που οφείλεται στις συνεχείς προσαρμογές που γίνονται σε ό,τι φορά τη χρηματοοικονομική υποστήριξη σε εθνικά συστήματα συγκέντρωσης στατιστικών δεδομένων. Μάλιστα, από την ε, εφαρμογή, από τους ρυθμούς εφαρμογής των πιστώσεων αυτών στα περασμένα χρόνια χρειάστηκε αυτή η προσαρμογή. Τώρα, για τον έλεγχο έχουμε μικρή μείωση 1,5%. Καταρχήν το 2013 δεν προβλέπεται υποστήριξη επενδύσεων σε σημαντικούς ελεκτικούς μηχανισμούς όπως είναι ε, σκάφη και πλοία περιπολίας γιατί αυτές είναι μεγάλες ε, δαπάνες και τώρα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του ελεκτικού κανονισμού, εκεί το μεγαλύτερο τμήμα του, των δαπανών έχει ήδη καλυφθεί από προηγούμενους προϋπολογισμούς. Για τον έλεγχο να πω τέλος ότι αυτό το κεφάλαιο ελέγχου περιλαμβάνει και τις επιδοτήσεις ε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου της Ελίας ε, που λειτουργεί στο Βίγκο και που είχε παγώσει ο προπολογισμό του στα επίπεδα του 2012 δυνάμει του βασικού κανόνα τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περιορισμό των διοικητικών δαπανών στο μέτρο του δυνατό φυσικά. Έρχομαι τώρα στο κεφάλαιο για τις ε, αγορές, τις ελευτικές αγορές. Ένα ζήτημα που ανέφερε ο κ. Ριβελίνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των μέτρων. Εδώ χρηματοδοτούμε κυρίως τα ίδια μέτρα σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις αγορών και τις ε, ιδιαίτερως απόκεντρες περιοχές. Υπάρχει μια μικρή μείωση σε σχέση με το 2012, μια ναι, και τα ποσά για τις ε, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμών είναι γύρω στα 20, ε, ε δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, επίσης, ελήφθη υπόψη ο ρυθμός ε, εφαρμογής τα περασμένα χρόνια, εξού και μερικές μειώσεις. Θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνοικης φυσικά τις εξελίξεις αγοράς, για να δούμε αν χρειάζονται περαιτέρω προσαρμογές και διορθώσεις. Τέλος, για την ε, πολιτική της θάλασσας, θαλάσσια πολιτική, δεν ε, απαιτήθηκαν αναλήψη υποχρεώσεων, ανάληψη υποχρεώσεων για το 2013 και αυτό εξηγείται από τη συμφωνία που είχε συναθεί επί του χρηματοπιστωτικού κανονισμού για το πρόγραμμα αυτό. Εκεί είχε αποφασιστεί ε, ένα front-loading για τις ε, πιστώσεις του προγράμματος για το 2011, ε, από τους προϋπολογισμούς του 2011 και του 2012. Οπότε, η αναλήψη υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στο, στα κονδύλια του προγράμματος αυτού περιλαμβάνονται στους προηγούμενους προϋπολογισμούς, ενώ οι δαπάνες εφαρμογής θα συνεχιστούν και το 2013. Και ζητήσαμε 50 εκατομμύρια ευρώ πιστώσεις πληρωμών για τις δράσεις του προγράμματος αυτό, Της θαλάσσης πολιτικής δηλαδή. Αυτά, εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να βρει μια ισορροπία στις προτάσεις για τον προϋπολογισμό του 2013 και να συνεχίσει τις πολιτικές της, αλλά ταυτόχρονα και να λάβει υπόψη την χαλεπή κατάσταση που δημιουργήθηκε από την κρίση για την Ευρώπη και για τους ε, πολίτες. Προσβλέπουμε σε συνέχιση της συζήτησης ε, στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο προϋπολογισμός του 2013. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Ριβελίνη. Εγώ γενικώ συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητού μας. Ε, από τότε που είμαι ευρωβουλευτής είχαμε περίπου ένα δις ε, ευρώ για, το, για την αλία. Φαίνεται ότι όλο και λιγότερα κονδύλια αφιερώνουμε στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Ενώ εξετάζουμε μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής το, η μείωση το 1,4% στο σύνολο της ανάληψης υποχρεώσεων είναι πολύ ε, πιο υψηλό από ό,τι περιμέναμε. Τώρα, με εξαίρεση το ΕΤΑ, το Ταμείο Αλληλείας και τη μείωση των διοικητικών δαπανών που είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα υπόλοιπα κεφάλαια διαπιστώνω πολύ σημαντικές μειώσεις. Στις αγορές έχουμε 11,7 στις αναλήψεις υποχρεώσεων, 10,9 μειώσεις στις πληρωμές, 11,03 διεθνές θέμα, 3,7 5,4 στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές. Το θέμα της διακυβέρνησης, στο οποίο υποδίδουμε τέτοια σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε 15,8% και 13,5% στις πληρωμές. Στο Ευρωπαϊκό Ταμείο φυσικά υπάρχει μια αναμενόμενη αύξηση, γιατί βρισκόμαστε στο τέλος τη περίοδου προγραμματισμού, οπότε είναι φυσιολογικό την τελευταία χρόνια να έχουμε περισσότερες δαπάνες. Στο θέμα της συντήρησης και πάλι έχουμε 4,3 και 5% στις πληρωμές. Στο θέμα του ελέγχου και δεν ξέρω γιατί αναφέρεται ότι αποφασιστήκε για το χρόνο να μην γίνουν επενδύσεις ούτε σε σκάφη ούτε σε ε, αεροσκάφη, αεροπλάνα περιπόλειες. Έχουμε ένα προπολογισμό με ένα δις. Πολύ λιγότερο δηλαδή από το Βαμβάκι ή άλλες χαζομάρες του Φεογκά και της Γεωργίας. Πραγματικά είναι δικαιολόγητος αυτός ο ισχνός προϋπολογισμός. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει ε, με το Συμβούλιο, γιατί μπορεί και εκεί να γίνουν περαιτέρω περικοπές. Αυτό είναι το σχέδιο προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν ώψη μια μεταρρύθμιση και δεδομένη τη κατάσταση στον τομέα, οι μειώσει, τον έλεγχο, τη συντήρηση, όλα αυτά τα θέματα είναι πραγματικά, τι να πω, άνω Σε ό,τι αφορά το Αλεκτικό οργανισμό. Μια χαρά πάει αυτό ο οργανισμό και εκεί κάνετε περίκοπέ. Δεν καταλαβαίνω Πώ τα δικαιολογείτε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να τα αναλύσουμε όλα περιπτωσιολογικά, να δούμε διεξοδικά το θέμα αναδημοσιονομική γραμμή για να δούμε αν όντω δικαιολογείται σε μερικέ περιπτώσει μείωση, αναλήψη υποχρεώσεων και πληρωμέ. Αλλιώ πραγματικά θα ενθάρρυνα τον εισηγητή μα να αναλάβουμε τι ευθύνε και να πάρουμε τι αποφάσει μα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριος Ρωμέβα και εγώ σύντομα. Νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η συζήτηση και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε μια κατάσταση που δείχνει ότι επενδύσεις, η έλλειψη επενδύσεων σε σημαντικά θέματα όπως ο έλεγχος δεν είναι, δεν είναι άμυρη συνεπειών. Εγώ θα, θα αναφέρω ένα παράδειγμα αυτής της εβδομάδας. Γνωρίζετε ότι άρχισαν, άρχισε η αλληλευτική περίοδος ε, για τα, τον αλλιευτικά γρηγρή και είχαμε ήδη καταγγελίες για πιθανές παραβιάσεις των ε, κανόνων της ΑΕΚΑΤ από το Παραγαδιάρικα και από τα γρηγρή. Δυστυχώς η απάντηση που μας έδωσε ο ελεκτικός οργανισμός είναι ότι δεν έχουν μέσα για να ε, διαλευκάνουν όλες τις καταγγελίες που λαμβάνουν. Οπότε, ενώ θέλουμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της ε, πολιτικής ελέγχου εφαρμόζοντας ε, τους κανόνες της ΑΕΚΑΤ στην συνεδρίαση του Νοεμβρίου, θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι γνωρίζαμε τι συνέβαινε, αλλά απλώς δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο για το συγκεκριμένο αλλιευτικό είδος. Έχουμε παράλληλα παραδείγματα και σε άλλα είδη αλίας. Και αν μειώσουμε τα ελάχιστα ούτως ή εργαλεία που έχουμε για έλεγχο και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες, πώς είναι δυνατόν ε, στη μετα... μετά τη μεταρρύθμιση να εξασφαλίσουμε σεβασμό των νέων διατάξεων. Νομίζω ότι στην αξιολόγηση της κατάστασης θα πρέπει να δούμε όχι μόνο ότι είναι αδικαιολόγητες μερικές μειώσεις, αλλά καταντούν και επικίνδυνες μερικές φορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώ εκ μέρου τη Εστέλ, διότι αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένη με προεκλογική εκστρατεία στη Γαλλία. Και θα είναι κρίμα για μα αν πάρει έδρα στο Κοινοβούλιο, θα είναι καλό για τη Γαλλία όμω. Μου είπε ότι η συνεργασία ανάμεσα στους κοιόδες και στους συζητητέ ήταν καλή και ότι εστάλει επιστολή στην Επιτροπή Περιπολογισμού. Από ό,τι ακούω είναι δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, να συνειδητοποιήσουμε ότι το Κοινοβούλιο ήδη το 2011 είπε πως θα ήταν αναγκαία μια αύξηση των πόρων για το ΕΤΘΑ σε σχέση με τα επίπεδα του 2013, για το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη να προτείνουμε πιστώσεις στα πλαίσια του νέου έτθα. Έπειτα, όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και η μεταρρύθμιση αυτή, όλη η μεταρρύθμιση, εξαρτάται από τη συλλογή δεδομένων. διότι πρέπει πάντα να, πρέπει να ξέρουμε πώς εξελίσσονται τα Από αποθέματα, χρειαζόμαστε αυτά τα επιστημονικά δεδομένα και τα χρειαζόμαστε πάντα και συνέχεια. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, αν δεν διαθέσουμε τους κατάλληλους πόρους για να γίνει σωστά αυτή η συλλογή δεδομένων, τότε όλη η μεταρρύθμιση κινδυνεύει να αποτύχει. Ο έλεγχος λοιπόν και η σωστή συλλογή δεδομένων είναι πράγματα που κοστίζουν χρήματα, αλλά πρέπει να τα πληρώσουμε. Δάλλος κινδυνεύει όλη η μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ. Muchas gracias. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Ο κύριος Ριβελίν. Grazie, Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς, όπως και οι συνάδελφοί μου, δεν είμαι διόλου ικανοποιημένος από την απόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προφανώ. όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει με την κρίση. Είναι κάτι το υπαρκτό. Όμως δεν μπορούμε να αρνηθούμε την πραγματικότητα κάνοντας κόλπα ε, με τα νούμερα και τους αριθμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί Κροατίας απέντησε ότι ίσως να λάβει μέρημνα στο μέλλον, αλλά για τις ε, θαλάσσιες πολιτικές, τις πολιτικές της θάλασσας, είπε ότι δεν προβλέπονται για την ώρα κονδύλια που μπορεί στο μέλλον να καλυφθούν με 12 εκατομμύρια ευρώ και δεν μας είπε πολύ τίποτε. Το επεσήμαναν όλοι οι συνάδελφοι, ιδίω ε, η κυρία Φράγκα, δεν μας είπε τίποτε για την αγορά αλίας. Εκεί η μείωση είναι πάνω από 10%. Είναι πραγματικά σημαντική. Επιπλέον, για τους ελέγχους παραδέχτηκε η Επιτροπή ότι οι περικοπές είναι επίσης σοβαρές. Προφανώς στην Ευρώπη ζούμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Όμως σε έναν τέτοιο τομέα δεν είναι λογικό να υπάρχουν τέτοια πλήγματα. Πέραν του κλάδου του βάμβακος ή του καπνού. Δεν αρκεί να μπερδεύει κανείς τους αριθμούς και να τους πηγαίνει από το ένα κεφάλαιο στο άλλο, πλήττοντας λίγο πολύ τους πάντες. Με ανησυχεί λοιπόν το μέλλον αυτού του τομέα. Με ανησυχεί γιατί έχουμε ευθύνη εναντί των συμπολιτών μας. Έχουμε ευθύνη εναντί των Ευρωπαίων εργαζομένων. Γνωρίζουμε ότι μπορεί να γνωρίσουμε μεγαλύτερες περικοπές ή μειώσεις. Θα φανεί και στην Ολομέλεια. Προς στιγμήν πάντως δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα φροντίσω να καταγράψω τα στοιχεία αυτά, να συντάξω ένα σχετικό κείμενο που να αντικατοπτρίζει την συζήτηση που μόλις κάναμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ριβελίνη. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη το υπαριθμό 16, που προβλέπει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Τον Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την έκθεσή της στα πλαίσια της Γενικής Πρότασης ε, για τις δημοσιονομικές προπτικές ε, και Ήδη ξεκίνησε η συζήτηση στη διάσκεψη των Προέδρων ε, ε, για ένα γενικό συντονισμό. Φαντάζομαι ότι καρπός του συντονισμού αυτού θα είναι μια διάμεση έκθεση που θα περιληφθεί ως παράρτημα στην έκθεση Επιτροπής και τον Ιούνιο, προς τα τέλη Ιουνίου, θα μας ε, ξαναενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Φερέιρα, για να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής του. Ευχαριστώ. Όλες οι ανησυχίες και προβληματισμός που ακούσαμε προηγουμένως από τους συναδέλφους εμφανίζονται και εδώ. Βέβαια τώρα δεν εξετάζουμε τον προϋπολογισμό του 2013, αλλά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα επηρεάσει όλους τους προϋπολογισμούς μέχρι το 2020. Οπότε όλες οι ανησυχίες που ακούσαμε προηγουμένως ε, έχουν λόγο ύπαρξης και μάλιστα ενισχυμένα και στη συζήτηση αυτή. Και στην έκθεση, στην, στο σχέδιο γνωμοδότησής μου προσπάθησα να λάβω υπόψη τις ε, ανησυχίες αυτές. Είπαμε στην αρχή πόσο σημαντικός είναι ο ελευτικός κλάδος και ότι αξίζει ιδιαίτερης προσοχής στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό το είχαμε πει επ' ευκαιρία και της προηγούμενης έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, έκθεσης Επιτροπής ΣΟΥΡ. Η έκθεση ΣΟΥΡ στην έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές τονίζει το σημαντικό ρόλο της αλίας Πέραν του, η πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 προβλέπει μια, ένα γενικό κονδύλιο 6 δισεκατομμυρίων, 685 εκατομμυρίων για την αλία και τις θαλάσσιες υποθέσεις συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσης και Αλίας, περισσότερα μετραγορά και κάποιες δαπάνες για τους περιφερειακούς οργανισμούς Έχουμε κατά μέσο όρο 955 εκατομμύρια για τον κάθε χρόνο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου του 2014-2020. Αυτό το ποσό, τα 955 ε, εκατομμύρια, είναι χαμηλότερα από, το, από τα 994 ευρώ που ήταν ε, ο μέσος όρος του προηγούμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, αυτό ελέγχθη υπόψη με την αριθμική αναπροσαρμογή. Κάτι που δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό και επισημαίνεται στην έκθεση. Πόλο δε μάλλον που κάποιοι στόχοι της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στρατηγική του 2020 για παράδειγμα να προωθηθεί η μετάβαση για, το, για ηλία με λιγότερο προϋπολογισμό για περιορισμένο αντίκτυπο της αλίας στα οικοσυστήματα, βιωσιμότητα των κοινοτήτων που εξαρτώνται από, από την παράκτη αλία και το θέμα της διαφοροποίησης. Όλοι αυτοί οι στόχοι που αναγκαίρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνοδεύονται από επαρκείς ε, πόρους για να υλοποιηθούν. Θα πρέπει λοιπόν το δημοσιονομικό πλαίσιο να ενισχυθεί, όχι να αποδυναμωθεί. Αλλιώ ε, κινδυνεύουμε να μην υλοποιήσουμε κανένα από αυτού του φιλόδοξου μεν απαραίτητου δε στόχου. Αυτή είναι μια ιδέα που αναφέρεται στη γνωμοδότηση. Μια άλλη ιδέα αφορά τον ε, ευάλωτο χαρακτήρα της ε, αλίας. Το νέο πολιτικό πλαίσιο προβλέπει για τη γεωργία που επίσης είναι ευάλωτο στην κρίση, μία σειρά μηχανισμών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Η γνωμοδότηση αναφέρει ότι ο ευάλωτος χαρακτήρας της γεωργίας θα πρέπει να ε, συγκριθεί με τον επίσης ευάλωτο χαρακτήρα της αλίας που επίσης υπόκειται στην κρίση, που επίσης υπόκειται σε αντίξωες καιρικές ηθίκες ή με μετεωρολογικές, ε, στις κλιματικές αλλαγές. Δεν είναι ε, δικαιολογείται λοιπόν γιατί να μην επεκτείνουμε τους μηχανισμούς αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτους ανάγκης της Γεωργίας και στην Αλία. Σε ό,τι αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Αυτό το ταμείο θα είναι ο βασικός μηχανισμός της ε, μελλοντική κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Θα πρέπει όμως να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα μέσα για να μπορεί να υλοποίηση του στόχου αυτής της κοινή αλληλευτική πολιτικής. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή του και επίση να γίνει μια προσπάθεια καλύτερου συντονισμού με του υπόλοιπου μηχανισμού της πολιτικής συνοχής. Τα θέματα απλούστευσης της πρόσβασης ε, στη χρηματοδότηση επίσης επισημένονται στην έκθεση. τονίζω ότι το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλία θα χρηματοδοτήσει και τομεί που αυτή τη στιγμή δεν με εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας που ισχύει σήμερα. Είναι πιο ευρύ το πεδίο του ΕΤΘΑ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλίας. Οπότε το μελλοντικό ταμείο θα πρέπει να έχει συμπληρωματικά κονδύλια, μια και θα χρηματοδοτήσει και νέου τομεί. Άρα χρειάζεται νέα μέσα, περισσότερα κονδύλια. Δεν μπορούμε να δεχθούμε η χρηματοδότηση των νέων τομέων να γίνουν ει βάρο ε, των ε, κονδυλίων που, που προβλέπονται για την αλία. Είναι μια άλλη σκέψη που α, ε, περιλαμβάνει η γνωμοδότηση. Θέματα όπως επιστημονική έρευνα στην αλία. Ένα θέμα που προβληματίζει την Επιτροπή γιατί δυστυχώς ε, δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά στοιχεία που ε, να οδηγούν σε μια διαχείριση της αλίας που θα στηρίζεται στη γνώση. Θα πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτηθούν περαιτέρω ε, επιστημονικές έρευνες για την αλία, το περιβάλλον και τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές για να καλυφθούν αυτά τα κενά που υπάρχουν στις γνώσεις μας στις επιστημονικές ως προς την αλία το θέμα της καλύτερης συγκέντρωσης ε, και διάθεσης των βιολογικών στοιχείων είναι ένα άλλο ζήτημα της γνωμοδότησης. Είδαμε ότι προτείνεται μείωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2013 στα θέματα αυτά. Οπότε θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό ο τομέας θα πρέπει να ληφθεί δόντω υπόψη στο επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Το θέμα τη ανάπτυξη τη υδατοκαλλιέργειας επίση είναι σημαντικό το θέμα των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της ε, ιδιαίτερης προσοχής που χρήζουν λόγω των ε, διαρθρωτικών μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν εξαιτία της γεωγραφικής τους θέσεις. θέσης. Επίσης, για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία υπάρχει μια παράγραφος το θέμα της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των Διεθνών Αλληλευτικών Συμφωνιών ε, τονίζεται και προτείνεται μία αλλαγή σε σχέση με το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας. Και ε, διατρανούμε και πάλι την απέτησή μας οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχουν ως παρατηρητές ισότιμα με τους εκπροσώπους των κρατών μελών σε όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης των διεθνών αλληλευτικών συμφωνιών δεδομένων των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των αλληλευτικών συμφωνιών. Αυτές είναι σε αδρές γραμμές ε, οι βασικές ε, προτάσεις της γνωμοδότησης. Υπάρχει και μία παράγραφος για την εξωτερική διάσταση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής αλλά προτιμώ να μην επεκταθώ στο σημείο αυτό. Αυτά προς το παρόν κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Φεραίρα. Θέλει το λόγο μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Όντω συνδέεται με την συζήτηση που μόλις κάναμε για τον υπολογισμό του 2013 διότι για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 έχουν τεθεί ε, φιλόδοξοι στόχοι μέσω της μεταρρύθμισης της κοινής ελληνικής πολιτικής για το Ταμείο της Θάλασσας και της Αλίας. Συμφωνούμε απολύτως με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να προβλεφθούν οι απαραίτητοι πόροι για αυτό το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και να στηρίξουμε την ε, μεταρρύθμιση της αλληλευτικής πολιτικής. Όντως, αυτό το ταμείο θα είναι βασικό εργαλείο για να στηρίξουμε και να επιδιώξουμε τους στόχους μας. Στα πλαίσια των συνολικών ποσών του Ταμείου, το σημερινό έτα πρικοδοτήθηκε με 4,3 δις ευρώ για το διάστημα 2007-2013. Το νέο ΕΤΘΑ που θα καλύπτει περισσότερα από το σημερινό ΕΤΑ πρικοδοτείται με 6,5 δις ευρώ. Άρα έχουμε λάβει υπόψη την επέκταση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου του στον υπολογισμό του ποσού για το 2014-2020. Επίσης, συμφωνούμε ότι απαιτείται απλούστευση για συγκεκριμένα μέτρα για την αλληλεία μέχρι κλίμακας και ότι πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την αλληλευτική επιστημονική γνώση. Αυτά έχουν ληφθεί υπόψη Στι προτάσει και για το Ταμείο και για την αλληλευτική πολιτική, την απλούστευση. Θα την πετύχουμε ενσωματώνοντα διαφορετικά προγράμματα υπό μια κοινή ομπρέλα, ένα κοινό ταμείο δηλαδή. Και συμπεριλαμβάνοντα το ΕΤΘΑ στο κοινό στατηγικό πλαίσιο με καταποκόπιν ποσά, την, κλίμακα, κλιμάκωση του κόστου και το καθεξή. Απλώ μια διευκρίνηση σε σχέση με το συνολικό ποσό που, με το οποίο προκοδοτείται το ΕΤΑ. Το μερίδιο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι το ίδιο όπως ισχύει για τις τωρινές δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Να αποσαφηνήσω ότι οι αριθμοί που έχουν υποβληθεί για το τμήμα αυτό, για τα θαλάσσια ζητήματα και την αλία και αυτά που αναφέρει η έκθεσή σας δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό. Εάν δούμε τις τρέχουσες τιμές, το συνολικό χαρτοφυλάκιο για την αλία και τις υποθέσεις είναι 7,5 δις πάνω από το επίπεδο των ε, αναλήψεων για το 2013 και από το 2015 και μετά. Οι δαπάνες λοιπόν για τις θελασσίες υποθέσεις και την αλία στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι πολύ κοντινέ κοντινές στις σημερινές, αυτές που ισχύουν με το παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν επίσης περισσότεροι συσχετισμοί μεταξύ του ΕΤΘΑ και του Ταμείου Συνοχής. Εδώ. Συνεχίζουμε να θεωρούμε το μεακό Ταμείο του ΕΤΘΑ που θα επιδιώκει τους στόχους μεταρρύθμισης του τομέα της αλίας. Για μας αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πηγαίνουν τα κοντέιλα και τα χρήματα εκεί που βρίσκονται οι αλείς, σε οποιαδήποτε περιοχή και αν βρίσκονται. Είτε σύγκληση είτε όχι. Και μια ακόμη μικρή διευκρίνηση. Φαίνεται ότι στην έκθεση έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι θα διακοπεί το πρόγραμμα για τι από κέντρε περιοχέ. Δεν ισχύει αυτό στην πρότασή μα. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε το ίδιο σύστημα με τι ίδιε περιοχέ και τα ίδια ποσά και στα πλαίσια του ΕΤΑ, του νέου μάλλον πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Συγγνώμη. Εδώ το διάστημα 2014-2020 δεν έχουμε αλλάξει την έμφαση που δίνεται στην μια περιοχή χρηματοδότησης ή δαπανών προς όφελος ή εις βάρος κάποιας άλλης. Ίσα ίσα που έχουμε την αίσθηση ότι οι στόχοι της μεταρρύθμισης της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής πρέπει να στηριχθούν επαρκώς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Δεν θέλει κανείς το λόγο. Οπότε περνάμε στο επόμενο σημείο, το Α, συγγνώμη, δεν σας πρόσεξα κύριε Φεραίρα. Έχω πρόβλημα με την όραση. President. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την πρόταση, αλλά πρώτα απ' όλα να κάνω ένα σχόλιο για τη σύγκριση μεταξύ του ισχύοντος ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας και του Μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλίας. Είπα στην αρχή και επιμένω ότι χρηματοδοτούν διαφορετικού τομεί Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και χρησιμο... χρηματοδοτεί τομεί που δεν εμπίπτουν σήμερα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελεία, αλλά χρηματοδοτούνται σήμερα από άλλου μηχανισμού, άλλου χρηματοδοτικού μηχανισμού που θα καταργηθούν όμω. Δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε απλώ μεταξύ των ποσών του ΕΤΑ, του Ταμείου Αλίας, και των μελλοντικών ποσών του ΕΤΘΑ, θάλασσας και αλίας γιατί έτσι δείχνουν, έχουμε, έχουμε μια υπεροχή του ΕΤΣΑ, αλλά μην ξεχνάτε ότι το ΕΤΣΑ θα χρηματοδοτήσει τομείς ε, που είναι πολύ πιο ευρύς από ότι οι τομείς του Ευρωπαϊκού Ταμείου ελίας, Σε ό,τι αφορά τώρα το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, όντως απαιτείται εδώ κάποια διευκρίνηση ώστε να αποφευθούν ε, παρερμηνίες στο εγγράφο. Στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020 προβλέπει 6 δισεκατομμύρια 685 εκατομμύρια ευρώ. Για το ΕΤΘΑ, ή μάλλον για το σύνολο, με τα μέτρα αγοράς, με, ε, τα, τα περιφερεια, τις περιφερειακές οργανώσεις αλλιές, κατά μέσο όρο 955 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο δηλαδή. Αυτό είναι ο μέσος ετήσιος όρος για την περίοδο 2014-2020. Για το 2013, αυτό που προβλέπεται με το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο, και νομίζω ότι οι τιμές αναφοράς ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το ίδιο έτος, σε σχέση με το 2011, είναι 984 εκατομμύρια. 984 είναι περισσότερο από 955. Έχουμε μία μείωση λοιπόν ε, του ετήσιου μέσου όρου για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, κάθε ετήσιο μέσο όρο είναι χαμηλότερο από τον ισχύοντα μέσο όρο του 2013, που είναι 984 εκατομμύρια. Θα πρέπει πάντως ε, να συμφωνήσουμε ως προς την ερμηνεία που δίνουμε της ανακοίνωσης ε, στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ως προς τον προϋπολογισμό προβλέπεται για το Ευρώπη 2020. Θα πρέπει λοιπόν να συντονίσουμε τις ερμηνείες μας και να μην ξεχνάμε ότι οι γενικές διαστάσεις του δημοσιονομικού πλαισίου, άσχετα με την αλία, ούτως ή άλλως παρουσιάζουν μια σχετική μείωση σε σχέση με το ισχύον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σχετική μείωση, σε ό,τι αφορά δηλαδή ποσοστό της, ε, του, ε, του ΑΕΠ. Οπότε αυτή η μείωση θα έχει μια αντανάκλαση σε όλες τις ε, δημοσιονομικές γραμμές και σε όλα τα κεφάλαια του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φερέρα. Οπότε περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, το σημείο 17, την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Είπαμε ότι θα συντάξουμε μια γνωμοδότηση επί της έκθεσης πρωτοβουλίας της Επιτροπής Ανάπτυξης. Την γνωμοδότηση αυτή την ανέλαβε και πάλι ο κύριος Ζωάν Φερέιρα. Α, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος, ξέχασα τη διορία για τις τροπολογίες για το σχέδιο γραμμοδότησης 11 Ιουνίου το μεσημέρι λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στη γνωμοδότηση Φερέιρα για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και τώρα ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Φερέιρα για να μα παρουσιάσει την επόμενη του γνωμοδότηση. Κύριε Λεβέν. Με συγχωρείτε. Κάτι μου διέφυγε. Ο Σολομό πότε θα συζητηθεί. Είναι το 15. Ε, Είπαμε ότι έγινε μια αντιστροφή των σημείων 15 και 21. Το 21 συζητήθηκε στη θέση του 15 και το 15 θα είναι το τελευταίο σημείο. Αυτό το είχαμε συμφωνήσει χθε όταν αλλάξαμε λίγο την ημερήσια διάταξη. Να δώσω το λόγο λοιπόν ε, στον κύριο Φερέιρα Δεν θα ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώ ας ακούσουμε, ακούσουμε πρώτα την παρουσίαση από την Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Uh, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή να παρουσιάσουμε την Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Συνοχή. Είναι η τρίτη έκθεση που δημοσιεύτηκε 15 Δεκεμβρίου του 2011. Αυτή η έκθεση ε, και δεν θα μπω στις ε, λεπτομέρειες τώρα γιατί είναι μια άσκηση που κάνουμε και ενδεχομένω να έχει επιπτώσεις και σε άλλους τομείς. Θα... Ε, περνάγαμε λοιπόν τρεις ώρες εάν συζητούσαμε όλες τις λεπτομέρειες. Απλά θα σας αναφέρω επιγραμματικά τη διαδικασία αυτή. Είναι μια έκθεση στην πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη που η Κομισιόν ετοιμάζει κάθε δύο χρόνια. Έχει λάβει την εντολή να το κάνει αυτό από το Συμβούλιο και κάνουμε εκθέσεις σχετικά με την ε, πρόοδο, πρόοδο συνοχής ε, για την ανάπτυξη, για πολιτικές και συμπεριλαμβάνεται και η Ελία στις εκθέσεις μας. Αυτές οι εκθέσεις συντάσσονται βασισμένες σε θεματικές συνεισφορές και από την Κομισιόν αλλά και από άλλα, άλλα όργανα και από τα κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν μια έκθεση αυτοαξιολόγησης τρόπον την Φέτος είναι μια κάπως πιο ε, σημαντική έκθεση διότι το 2011, μάλλον διότι η έκθεση του 2011 θα ακολουθηθεί από μια πρώτη έκθεση του Κοινοβουλίου για την πολιτική συνοχή και την ανάπτυξη που θα γίνει από την κυρία Γιάστραμ της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Είχαμε σημαντικές συνεισφορές από μέρους της που θα κάνει την επόμενη μας έκθεση για το 2013 ακόμα καλύτερη. Το έγγραφο εργασία τη Κομισιόν αποτελείται από την έκθεση, δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και η έκθεση αυτή καλύπτει την περίοδο από το 2009 ως το 2011. Σε αυτή την έκθεση επικεντρωθήκαμε σε πέντε προκλήσεις που αποφασίστηκαν μετά από την έκθεση του 2009 ε, μπορεί και τα δημοσιονομικά, η κλιματική αλλαγή και η αλληλεία συμπεριλαμβάνεται σε αυτά η μετανάστευση και η ασφάλεια. Επίση υπάρχει μια, ε, ένας άλλος τομέας που αναφέρεται στην πρόοδο και των ειρηνευτικών στην πρόοδο γενικά για τα κρατη και για την Κομισιόν. Διαιρείται σε τρία ε, μέρη. Πρώτον, τα γενικά ε, θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Ε, αναφέρονται οι δομές, για την πολιτική συνοχή, η χάραξη πολιτικής για την ανάπτυξη. Ε, αυτά συντάσσονται από ομάδες, περνάνε από διαφορετικές ομάδες, μετά από συμβουλευτικές διαδικασίες. Φυσικά η, ο δεύτερος τομέας της έκθεσης καλύπτει τις πέντε προκλήσεις που ανέφερα πιο πριν. Ε, ε, αυτό που σα ενδιαφέρει εσά είναι οι, ο για την ασφα... ασφάλεια, όπου αναφέρεται και το τομέα της αλληλεία. Τα τελευταία δύο χρόνια φυσικά έπρεπε να θέσουμε τις προτεραιότητές μας στην έκθεση. Επικεντρωθήκαμε στα μεγάλα ζητήματα, στους μεγάλους φακέλους. Η μεταρρύθμιση της αλληλευτικής πολιτικής ήταν ένας από αυτούς. Ε, και το είδαμε από την πλευρά της ανάπτυξης. Τι υπάρχει στην πρόταση λοιπόν για την μεταρρύθμιση και τι πρόοδο έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε στον τομέα της χρηματοδότησης. Η δομή ε, συμφωνήθηκε το 2009, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια ο τομέας της αλίας δεν μπορεί να γίνει ξεχωριστό τομέα στην έκθεση ανάλογα με τις συγκυρίες. Μπορεί να αλλάξει λοιπόν στο μέλλον. Το τρίτο σημείο της έκθεσης αναφέρει μερικά από τα μαθήματα που έχουμε διδαχθεί και τις επόμενες προκλήσεις για το μέλος που εντόπισαν τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας πιστήσω την προσοχή στην επόμενη έκθεση, στο follow-up του φακέλου. Η σύνταξη της έκθεσης έδειξε την ανάγκη για στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία, για την συνοχή και την ανάπτυξη. Περισσότερη συνεργασία, λιγότερη, λιγότερη ατομική εργασία, συνεργασία των ε, θεσμικών οργάνων μαζί με τα κράτη-μέλη, OECD Καθώς και σε διεθνείς ε, διαδικτυακές πλατφόρμες. Είναι μια ιδιαίτερη μορφή έκθεσης, διότι δεν αναφέρεται μόνο σε δράσεις. Έχουμε βέβαια ακόμα κενά, γιατί είναι μόλις η τρίτη μας έκθεση. Γι' αυτό λοιπόν και είναι ευπρόσδεκτα οποιαδήποτε σχόλια και οποιασδήποτε προτάσεις για βελτίωση. Τέλος, μέτρα που λάβαμε τα τελευταία χρόνια ο έλεγχο, η συλλογή δεδομένων και η χωρητικότητα της συλλογής δεδομένων πρέπει να ενισχυθούν έτσι, σε πολλούς τομεί, συμπεριλαμβανομένης και τη αλληλεία, έτσι ώστε να συλλέξουμε στοιχεία επαρκή για σωστή επεξεργασία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί είμαι σίγουρη ότι το έχετε συζητήσει εκτενώς μια και είναι ο τομέα σας. Θα περάσω όμως σε αυτά που σκοπεύουμε να κάνουμε για τον επόμενο χρόνο. Ήδη έχουν γίνει ορισμένε συζητήσει στην Επιτροπή ανάπτυξη στην αρχή του χρόνου για την έκθεση. Ε, θα έχουμε συνεισφορέ από πολλές επιτροπές Συμπεριλαμβανομένε τη έκθεση της κυρίας Γιάστραμ και πραγματικά ε, περιμένουμε από, από εσά και από τη δική σας έκθεση περισσότερη συμβολή, μεγαλύτερη συμβολή και βοήθεια για το τι ε, μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Διότι η φωνή του Κοινοβουλίου δεν έχει ακουστεί αρκετά. Δεν έχει παρατηρηθεί μεγάλη συνεισφορά. Συμπεράσματα τώρα της έκθεσης στις 14 Μαΐου του 2012 κάναμε σύσταση στο Συμβούλιο να συνεχίσει τη δουλειά του και να ενισχύσει την, ε, τις προσπάθειες για ε, την πολιτική συνοχής για την ανάπτυξη αλλά και τα ίδια τα κράτη-μέλη. Στα κράτη-μέλη συστάθηκε να συμμετέχουν και εκείνα και να ενισχύσουν και εκείνα τις ε, δικές τους προσπάθειες. Αυτή είναι μία από τις προκλήσεις μας για τα επόμενα χρόνια, μία αρκετά μεγάλη πρόκληση θα έλεγα. Δεν θα πω στα ψηλά γράμματα της έκθεσης για να μην πλήξετε. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φερέρα τώρα. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο σύντομα σχόλια. Πρώτον, να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μα που μια τέτοια έκθεση, που είναι μια σημαντική έκθεση όπω είπε και η πρόσωπο τη Επιτροπή, αξιολογώντας τη συνοχή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ανάπτυξης, δεν διατίθεται στις επίσημες γλώσσες. Αυτή είναι η πρώτη μου σημείωση και επικριτικό σχόλιο. Ένα τόσο σημαντικό έγγραφο θα πρέπει να διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Εκ όσων γνωρίζω, διατίθεται μόνο στα αγγλικά και η Επιτροπή Κάτι θα έπρεπε να κάνει ώστε να προσυντομότερα, ώστε να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Να μεταφραστεί και στις 23 επίσημες γλώσσες. Μια δεύτερη παρατήρηση για να πω ότι έχω την αίσθηση ότι εμείς ως Επιτροπή Αλίας έχουμε αναλάβει ακριβώς μια έκθεση για το θέμα αυτό, την συνοχή των ευρωπαϊκών πολιτικών σε σχέση με την ανάπτυξη και ακριβώς έχουμε εδώ και δύο δεκαετίες τουλάχιστον ε, συμφωνίες με τρίτες χώρες που είναι αναπτυσσόμενες χώρες. Εδώ και 20 χρόνια το λιγότερο υπάρχει και διάσταση της συνεργασίας στις συμφωνίες αυτές. Δηλαδή τουλάχιστον 20 χρόνια τώρα ε, αντί να δίνουμε απλώ κονδύλια στι χώρε αυτέ ε, με αντάλλαγμα να εκμεταλλευόμαστε του φυσικού ε, πόρου του, θα έπρεπε να του δώσουμε και κάποια κονδύλια ώστε να μπορέσουν να απτύξουν οι ίδιοι αυτού του φυσικού πόρου, του αλληλευτικού. Θα έπρεπε να μπορούν δηλαδή τα αλληλευτικά του αποθέματα εκείνοι να τα αξιοποιούν και μετά να τα εξάγουν με την προστιθέμενη αξία που του αναλογεί. Αυτό θα ήταν το θετικό αποτέλεσμα για αυτέ τι χώρε. Τώρα, 20 χρόνια αργότερα, βλέπουμε πόσες ελλείψεις έχει αυτή η διάσταση της συνεργασίας μέσα από αλληλευτικές συμφωνίες. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία. Το βλέπουμε μέσα από την έκθεση για την συνοχή σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή πολιτική. Τι πήγε άσχημα με την αλληλευτική πολιτική. Αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σήμερα τα κονδύλια που αναγνωρίζοντας τους διάφορους τομείς είναι ελλειπή προκειμένου να πετύχουμε τους επιδιωκόμενους στόχους. Τι πρέπει να αλλάξει λοιπόν στον τομέα αυτό για να είναι πιο αποτελεσματική η τομεακή προσέγγιση. Η απόδοση κονδυλίων στις τρίτες χώρες, η συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Φερέιρα για την εισαγωγή του αυτή. Ωστόσο, ε, είμαι κάπως απογοητευμένη από την παρουσίαση της Κομισιόν, διότι όπως είπε και ο κύριος Φερέιρα, η έκθεση αυτή ε, δεν είναι σε όλες τις επίσημες γλώσσες, ε, γίνεται μόνο κάθε δύο χρόνια, είναι εξαιρετικά σημαντική Διάβασα το έγγραφο εργασίας της κυρίας Γιάστραμ, της εισηγήτριας για, για την πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη και οι περιοχές οι περιοχές που επηρεάζουν περισσότερο Συγγνώμη, διαβάζω από τα Σουηδικά, θα προσπαθήσω να μεταφράσω. στι αναπτυσσόμενες χώρες, λοιπόν, είναι η εμπορική πολιτική, η αγροτική πολιτική και η ελευθερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν περιμένω να ακούσω από την Επιτροπή ποια είναι τα συμπεράσματα στην ε, συνοχή της πολιτικής και την ε, πολιτική για την ανάπτυξη. Αυτό θα με ενδιέφερε. Διότι, όπως είπα και ο κύριος Φεραίρα, αυτή η πολιτική λαμβάνει χώρα εδώ και 20 χρόνια και τα συμπεράσματα από την Κομισιόν θα ήταν πολύ χρήσιμα. Παρακολουθώ το ζήτημα στενά και θα ήθελα να το συζητήσω και περαιτέρω. Εάν η Κομισιόν δεν θέλει να μπει σε λεπτομέρειες, ε, εγώ πάντως δεν θα βαριόμουν καθόλου να ακούσω τις λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε κύριε Λοβέν. Θέλει άλλος κανείς το λόγο. Θέλει να πει κάτι καινούργια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια στιγμή πρώτα κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ. Εγώ διάβασα την έκθεση της Επιτροπής και τουλάχιστον η σύνοψη της έκθεσης δίνει την εντύπωση ότι κάνει μια σχετικά επιφανειακή επισκόπηση, κάπως αφιψηλού της κατάστασης και δεν καταλαβαίνω και μερικές διαπιστώσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει ότι προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, λέει ότι η διαπραγμάτευση για τις ελληνικές συμφωνίες θα πρέπει να στηρίζεται στις προτεραιότητες του συμβαλόμενου μέρους προκειμένου να εξασφαλιστεί κατάλληλη ανάπτυξη της, αληφ... του κράτους και της οικονομίας του γενικά. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθήσει τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών. Αυτό που διαπιστώνουμε όμως, και το είπαμε και χθε στους εκπροσώπους της Επιτροπής, είναι ότι ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και των τρίτων χωρών, ε, αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα στη σύναψη συμφωνιών, γιατί τα συμφέροντα των τρίτων χωρών αλλάζουν Και αντί να εστερνιστούν ε, τα κριτήρια και τις αρχές μας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το σεβασμό, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική προστασία, αυτό που διεκδικούν οι τρίτες χώρες είναι συμφωνίες ανεφόρων. Για παράδειγμα με την Κίνα. Τους δίνουμε περισσότερα κονδύλια, ε, τους ε, υποβάλλουμε περισσότερους όρους και έτσι τους δίνουμε πάτημα για να μην υπογράφουν συμφωνίες. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω αυτή την αντίφαση και να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ανάλυση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής, λάβατε υπόψη τις αλληλευτικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες. Γιατί δεν εξαρτώνται όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι όλα στα δικά μας χέρια. Μπορεί πριν από 20 χρόνια να ίσχυε αυτό, αλλά τώρα πια δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι εξαρτάται από εμά και αν εμείς επιλέξουμε μια συμφωνία θα ευοδοθεί και όλα. Εσείς ε, δεν τη διαπιστώνετε αυτή την αντίφαση και πώς θα εξασφαλίσουμε τη συνοχή, την ε, επιθυμητή συνοχή και πώς θα περιλάβουμε αυτές τις αναδυόμενες οικονομίες σε συστήματα γενικευμένων προτιμήσεων, αφού πρόκειται για αναδυόμενες οικονομίες. Πού βλέπετε τη συνοχή εδώ με την αναπτυξιακή πολιτική. Παρακαλώ να δώσει μια απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω όμως όσον αφορά την διαθεσιμότητα της έκθεσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Δεν το έχουμε κάνει για λόγους οικονομίας. Η έκθεση συντάσσεται κάθε δύο χρόνια, ορισμένα μέρη της επαναλαμβάνονται και εμείς διατηρήσαμε το μορφότυπο του εγγράφου εργασίας που ε, είναι σε μία από τις γλώσσες εργασίας της Κομισιόν, μία από τις τρεις. Προς το παρόν είναι μόνο διαθέσιμο στα αγγλικά. Όσον αφορά για την αλληλεία και για την συνεργασία τώρα. Δεν θέλω να σας δώσω ελπίδες για την ίδια την έκθεση, διότι η έκθεση ως ε, άσκηση ε, είχαμε την εντολή να μην κάνουμε προπάσεις, προτάσεις. Διότι τότε δεν θα ήταν έκθεση. Υπάρχουν άλλα είδη κειμένων που κάνουν προτάσεις. Αυτό ήταν μια άσκηση, μια έκθεση για να αποτυπώσουμε τις πολιτικές έτσι όπως ήταν τη συγκεκριμένη στιγμή. Γι' αυτό και υπάρχουν αντιφάσεις στην έκθεση και ίσως αυτό ε, θέλετε να πείτε τώρα. Περιγράφουμε τις πολιτικές όπως, έχουν αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να δούμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αλλά φυσικά δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, γι' αυτό και θέλουμε να συνεχίσουμε. Δεν είναι όμως αντικείμενο της έκθεσης να προτείνει μεγάλες και καλές λύσεις, δεν είναι αυτό το αντικείμενο. Και προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτό. Δεν θα τώρα μπω σε λεπτομέρειες, θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου. Oui, si vous le permettez, je vais compléter les, les propos de... Εάν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω τα όσα είπε η συνάδελφος, εγώ παραμένω εξ ονόματο τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ και να κάνω και εγώ κάποιε παρατηρήσει. Το πρόβλημα που έχουμε στι περισσότερε χώρε εταίρου ή δικαιούχου των διμερών συμφωνιών αλεία είναι ότι το τομέα αλεία δεν λαμβάνεται υπόψη ε, στον προγραμματισμό τη αναπτυξιακή πολιτική του ω προτεραιότητα. Κάποιε ορίζουν προτεραιότητα την υγεία, την οδοποιία, τα σχολεία. Υπάρχουν βεβαίω εξαιρέσει όπως τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού. Όμως ο τομέας της αλληλείας δεν θεωρείται προτεραιότητα. Αυτό είναι ένα πρώτο πρόβλημα. Όταν έχουμε λοιπόν μια αλληλευτική συμφωνία, διμερή, υπάρχει ε, ένα σκέλος ε, τομεακής στήριξης το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί ως παρότρινση, ώστε η αναπτυξιακή πολιτική να είναι συνεκτική και να συμπληρώνει τη δική μας δράση με επενδύσεις στον τομέα της αλίας. Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντοτε. Διότι καταλήγουμε στο αντίστροφο. Λέμε, α, υπάρχει αλληλευτική συμφωνία, χρηματοδοτεί διευθυντικέ ε, αλλαγέ στον τομέα τη αλεία, άρα δεν θα ασχοληθεί με αυτό η πολιτική αλεία. Ένα δεύτερο πρόβλημα λοιπόν υπάρχει εδώ τελικά όχι συμπληρωματικότητα, αλλά διαχωρισμό των τομέων. Και να αντιδράσω και στο σχόλιο ότι η τομεακή στήριξη αυτό το σκέλος έχει αποτύχει ως τώρα. Συγγνώμη, αλλά εδώ θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό στη διαπίστωση. Βεβαίως υπάρχει έλλειψη πληροφοριών ή ενημέρωση για το τι χρηματοδοτείτε, τι στηρίζετε στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών. Όμω μπορώ να σα βεβαιώσω ότι στο σύνολο των συμφωνιών τα πράγματα πάνε μάλλον καλά. Υπάρχει μια σειρά από ενέργειε για τη διακυβέρνηση τη Αλία. Δεν είναι τόσο ορατέ, όμω πολλά χρηματοδοτούνται για την παρακολούθηση λόγω χάρη των θαλάσσιων γεωγραφικών περιοχών των ζωνών για την ενίσχυση των επιστημονικών δυνατοτήτων αυτών των χωρών, για την συμμετοχή του σε περιφερειακούς οργανισμούς αλίας. Οι ενέργειε αυτέ δεν είναι θεαματικέ, δεν είναι φαντασμαγωρικέ. Δεν αφορούν φυσικέ εγκαταστάσει, ε, λιμάνια ή εγκαταστάσει των λιμένων. Είναι περιορισμένα. Όντω, το είπε ο κ. φεραιρα Φεραίρα, έχουμε 200-300 ευρώ πολλέ φορέ στα χέρια μα. Δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακρύτερα. Μπορούμε να στηρίξουμε κάπως την διακυβέρνηση, να δώσουμε κάποια διοικητική αρρωγή στον τομέα της αλληλεία της χώρας αυτές, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και επαναστατικέ ή ριζοσπαστικέ αλλαγές ή παρεμβάσεις. Το τμήμα λοιπόν που αναλογεί στην τομεακή στήριξη πάει καλά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία των ίδιων των χωρών και θα πρέπει αυτό να είναι συμπλήρωμα στην αλληλευτική του δραστηριότητα. Ιδάλω, ξεφεύγουμε από τον τομέα της αλίας και περνάμε στον τομέα της ανάπτυξης. Όμως αυτές οι αλληλευτικές συμφωνίες δεν είναι εργαλεία αναπτυξιακά, είναι μέρος της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ευχαριστούμε κύριε Λόβεν. Ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο. δεν φανταζόμουν ότι η έκθεση συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής θα υπέβαλε και συστάσεις. Περιμένω αξιολόγηση. Βλέπω όμω ότι ξαναπαίρνει το λόγο Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Προσπαθεί να μα το ξαναεξηγήσει. Μα η ιδέα τη συνοχή αναπτυξιακή πολιτική είναι να πάρουμε μια απόσταση, να κάνουμε μια επισκόπηση των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε κατά πόσο είναι συνεπεί με, με του αναπτυξιακού μα στόχου. Αυτή την αξιολόγηση θα πρέπει να την κάνετε και να συνεννοηθείτε πριν έρθετε να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ κύριο Φεραίρα για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να τονίσω αυτά που είπε η κυρία Λόβεν. Η διάσταση της ε, ε, συνεργασίας ή της τομεακής υποστήριξης ε, σε περίπτωση που χαρακτηριστεί από δεν σημαίνει ότι δεν έγινε απολύτω τίποτα σε κανένα τομέα. Αυτή η διαπίστωση της γενικής αποτυχίας ξεκινά από την αναγνώριση ότι από την άποψη των μεγαλεπίβολων στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής, δηλαδή από, την, τον περιορισμό της εξάρτησης των χωρών, από το να καταστούν δυνατές να εκμεταλλεύονται μόνοι τους, ε, τις, ε, τους τις ε, τους πόρους, αντί να ανοίγουν την εκμετάλλευση της Ευρωπαϊκής Ένωση. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρείται αποτυχημένη η αναπτυξιακή πολιτική. Πέρυσι στείλαμε αποστολή της ε, Επιτροπής μας στην Μαυριτανία. 700 χιλιόμετρα ακτές έχει η Μαυριτανία, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα λιμάνι εκφόρτωσης ελευτικών προϊόντων. Και η χώρα αυτή εδώ και 20 χρόνια συνάπτει ελευτικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά, που προβλέπει και αναπτυξιακό σκέλος. Ενίσχυση τη ανάπτυξη του αλληλευτικού κλάδου της ε, 20 ολόκληρα χρόνια δεν μπόρεσαν να κατασκευάσουν ούτε ένα λιμάνι ε, καταστάσεις εκφόρτωσης μέσα σε 700 χιλιόμετρα ακτέ, Από τη στιγμή που δεν μπορεί κανένα να ε, αποπλέψει και να εκφορτώσει ε, αλλιεύματα στη Μαυριτανία, η προστιθέμενη αξία της εκφόρτωσης ε, εκτοπίζεται εκτός της Μαυριτανίας Από αυτή την άποψη, η αναπτυξιακή προσπάθεια ήταν αποτυχία. Γιατί δεν κάναμε λιγότερο εξαρτημένε αυτές τις χώρες Γιατί οι αλληλευτικές συμφωνίε ούτε τομεακή υποστήριξη παρήχαν, ούτε μείωσαν την εξάρτηση των χωρών αυτών από την αναπτυξιακή βοήθεια. Άρα, όντω, υπήρχε αποτυχία από αυτή την άποψη. Και δεν περιορίζεται το θέμα μόνο στι αλληλευτικές συμφωνίες είναι γενικό πρόβλημα της πολιτικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, οι ελευτικές συμφωνίες αποτελούν ένα τμήμα μόνο της ευρύτερης πολιτικής συνεργασίας και στην έκθεση αυτή ουσιαστικά μιλάμε για τη γενικότερη πολιτική της ε, συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Και αυτή την άποψη η ανεπάρκεια της αναπτυξιακής πολιτικής, ε, η αποτυχία της μερικές φορές ως προς τις αλληλευτικές συμφωνίες ε, θα πρέπει να αναγνωριστεί. Καλώς. Περνάμε στο επόμενο σημείο τώρα, το σημείο 18, τη θέσπιση του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, Ορίζω 2020. Το Δεκέμβριο αποφασίσαμε να συντάξουμε γνωμοδότηση επί της έκθεσης ουσίας της Επιτροπής Βιομηχανίας. Την γνωμοδότηση την ανέλαβε ο κύριος Τσουκαλάς, στον οποίο και δίνουμε το λόγο για την ανταλλαγή απόψεων. Έχετε το λόγο κύριε Τσουκαλά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα σήμερα να σας εκθέσω τις, τον βασικό πυρήνα των σκέψεών μου για την υποκατάθεση γνωμοδότηση η οποία θα πρέπει να παρουσιαστεί στις αρχές Ιουλίου. Άκουσα με μεγάλη ευχαρίστηση προηγουμένως να αναφέρεται συχνά η έρευνα και η καινοτομία στη συζήτηση για την αλληλεία. Ο Ρίζων 2020 περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, το οποίο έχει έναν αρχικό προϋπολογισμό 82 δισεκατομμυρίων Υποτίθεται ότι τα 82 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι περισσότερα από τα 54 του 7 πλαισίου, αποτελούν μια μεγάλη πρόοδο σε σχέση με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ορίζοντα 2020. Ο κύριος Έλερ, ο οποίος διευθύνει τις συζητήσεις οριζόντια για τη σύνταξη των αναφορών σχετικά με τον ορίζοντα 2020 διαφόρων επιτροπών έχει καταλήξει το συμπέρασμα ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι ονομαστικά μόνο τόσο μεγάλος το, ο αριθμός είναι ενδεικτικός και πιθανότατα δεν πρόκειται να μείνει εκεί. Υπολογίζει ότι είναι περίπου μια αύξηση 6 έως 7%. Σας λέω αυτό το γενικό περίγραμμα για να έχετε υπόψη σας πώς ακριβώς αρχίζει και διαμορφώνεται το κλίμα σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετικά τώρα με την έρευνα και την καινοτομία στην, στον τομέα ευθύνης της Επιτροπής μας, δηλαδή την Αλία, θα ήθελα πρώτα να σας πω, μολονότι ίσως να είναι ε, κοινότοπα το, αυτό που θα πω για σας εδώ στην Επιτροπή Ελίας, όμως πρέπει να στηρίξω ε, για ποιο λόγο η έρευνα και η καινοτομία στην Αλία είναι σημαντική, πού στηρίζω αυτή μου την άποψη και ποιες νομίζω ότι θα πρέπει να είναι οι προτάσεις της Επιτροπής μας για να συμπεριληφθούν στον ορίζοντα 2020. Άκουσα τον κύριο Φερέιρα πριν να λέει για 800 χιλιόμετρα ακτογραμμής οι συνολικές ακτογραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 68.000 χιλιόμετρα, αφορούν 22 κράτη-μέλη και περίπου το 50% των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοικούν σε απόσταση μικρότερη από 50 χιλιόμετρα από την ακτή. 5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ασχολούνται σχετικά με τη θάλασσα θέσεις εργασίας και προσφέρουν πάνω από το 5% του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θαλάσσια, τα υδάτινα περιβάλλοντα και οι σχετικές δραστηριότητες είναι απαραίτητα για την ευρωπαϊκή κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Ο ρόλος του θαλασσίου περιβάλλοντος γίνεται ακόμα πιο σημαντικός αν αναλογιστούμε τη σημασία και τις δυνατότητες του στην αντιμετώπιση των συγχρόνων προκλήσεων, όπως είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα, η κλιματική αλλαγή, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η υγεία, η αύξηση του πληθυσμού που θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση ζήτησης τροφίμων και αλλιευμάτων συνεπώς. Η αλληλεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το θαλάσσιο περιβάλλον καθιστά αναγκαία τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα, καθώς συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης αλληλείας, η οποία θα σέβεται το περιβάλλον και ταυτόχρονα θα λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και οι οικονομικές ανάγκες των παρακτήων και νησιωτικών κοινοτήτων. Μέχρι και σήμερα, πάνω από το 90% της θαλάσσιας βιοπικιλότητας παραμένει ανεξέταστο και αυτή η έλλειψη αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων για την οποία μίλησε και ο κύριος Γκάλαχερ καθιστά τις προσπάθειες για την επίτευξη αηφόρου διαχείρισης των αλλιευτικών αποθεμάτων των ευρωπαϊκών θαλασσών ακόμα πιο δύσκολες. Στο τρέχο πρόγραμμα έρευνα, το 7ο πλαίσιο, ο ετήσιος προϋπολογισμός που διατίθεται για τους κλάδους της αλληλείας, τη υδατοκαλλιέργειας και της θαλάσσιας βιοτεχνολογίας είναι περίπου 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. 30 εκατομμύρια ευρώ για αλληλεία και υδατοκαλλιέργεια και 20 για θαλάσσια βιοτεχνολογία ποσό που μπορεί να φαίνεται σημαντικό, αλλά φαίνεται από το αποτέλεσμα ότι δεν είναι επαρκές. Δεδομένης της αύξηση του προϋπολογισμού θα πρέπει συνεπώς να επιτευχθεί και αύξηση πρέπει να αυξήσουμε το ποσό που προβλέπεται για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα. Οι κύριε σκέψεις μου σχετικά με το report το οποίο πρόκειται να σας καταθέσω θα επικεντρωθούν κυρίως στα εξής σημεία. Πρώτον, τη σημασία και τη συμβολή της έρευνας στις θαλάσσιες και ναυτιλιακές δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των συγχρόνων κοινωνικών προκλήσεων μέσω της διατομεακής προσέγγισης. Την στενότερη συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς μια ουσιαστικότερη συνεργασία των ερευνητικών προγραμμάτων με τα διαρθρωτικά προγράμματα θα είχε θετικά αποτελέσματα στον τομέα της αλληλείας. Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνητών και ατόμων που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τον κλάδο, εκπρόσωποι του ελευτικού τομέα, επιχειρήσεις, καταναλωτές, φορείς χάραξης πολιτικής. Ο αλληλευτικός κλάδος πολλές φορές θεωρεί την έρευνα ως εμπόδιο για την αλληλευτική δραστηριότητα και αυτή η αντίληψη θα πρέπει να αλλάξει. Σχετικά με τον προϋπολογισμό, θετικό είναι το γεγονός ότι η έρευνα στον τομέα της θαλάσσιας και της, της θάλασσας και της ναυτιλίας έχει συμπεριληφθεί ρητά στον ορίζοντα 2020. Είναι το τμήμα 3 της κοινωνικές προκλήσεις και διευκολύνει με τον τρόπο αυτό τις διατομεακές δράσεις στον τομέα της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας για τις μελλοντικές δραστηριότητες. Ωστόσο, Υπάρχει ακόμα η ανάγκη να ενισχυθεί εν λόγω έρευνα με επαρκέστερη χρηματοδότηση. Χωρί τα κατάλληλα κονδύλια, το μεγάλο δυναμικό των θαλασσίων επιστημών και τη τεχνολογία του τομέα θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Αυτέ είναι κάποιε ιδέε που σκέφτομαι να αναφέρω στην γνωμοδότησή μου. Με χαρά περιμένω τα σχόλια και τι σκέψει σα, ώστε η Επιτροπή μα να παρουσιάσει ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο κείμενο που θα ανταποκρίνεται στι ανάγκε της σύγχρονης εποχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσουκαλά. Το λόγο τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά θα ακούσουμε τους συναδέλφους. Παρακαλώ. Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τα πολύ χρήσιμα σχόλια που μόλις έγιναν και τα γενικά σχόλια τα οποία σκοπεύετε να κάνετε. Πιστεύω ότι τα περισσότερα σημεία που θίξατε και συμφωνώ ότι δεν είναι λεπτομερή σε αυτό το στάδιο, όμως σίγουρα ελπίζουμε να βρούμε τρόπο να επιτύχουμε συνοχή με τα διαρθρωτικά ταμεία. Υπάρχει λοιπόν, ε, έχουμε μεγάλη προοπτική με τη συνεργασία ε, με άλλες πηγές από ευρωπαϊκά ταμεία. Φυσικά αυτό απαιτεί οι επιμέρους περιφέρειες να εναρμονίσουν τις δραστηριότητές τους έτσι ώστε να συμπίπτουν και με τις ε, δικές σας. Οπωσδήποτε σκοπεύουμε να αυξήσουμε τον προπολογισμό. Η Κομισιόν έχει προτείνει μια σημαντική αύξηση, όπως είπατε και εσείς, ε, για το γενικό πακέτο για την έρευνα και συγκεκριμένα για την βιοοικονομία, το οποίο συμπεριλαμβάνει την αλληλεία, την γεωργία και την ε, θαλάσσια τεχνολογία. Ε, θα διπλασιάσουμε την χρηματοδότηση. Αυτό προτείναμε. Φυσικά αυτό είναι πρόταση και δεν είναι ακόμα εγγυημένο. Εξαρτάται από άλλους παράγοντες. Τουλάχιστον όμως η Επιτροπή έχει δείξει προθυμία και έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά αναγνωρίζοντας την σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα αυτό. Υπογραμμίσατε την πολυτομεακή προσέγγιση και εμείς σίγουρα αρχίσαμε να το κάνουμε αυτό κατά από το πρόγραμμα πλαίσιο 7 με τις, ε, για αρκετά ε, θέματα. Προσπαθήσαμε, για παράδειγμα, τον τομέα του περιβάλλοντος ε, να τον εντάξουμε την υδατοκαλλιέργεια, την θαλάσσια βιοτεχνολογία, να τα συνδέσουμε με τους τομείς ε, των μεταφορών και της ενέργειας και σίγουρα ε, είχαμε κάποιες επιτυχίες στα πρώτα στάδια του προγράμματος. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε, να πάμε πιο πέρα στα επόμενα, ε, στα επόμενα πακέτα μετά το 2020 με την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχουν και τα κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτούς τους τομείς. Όλο το πρόγραμμα πλαίσιο, θα ήθελα να πω, όλο το νέο πακέτο που θα έρθει το 2020 θα ενώσει όχι, ε, όχι μόνο την, ε, τις ε, δραστηριότητες έρευνες, αλλά και ένα σημαντικό μέρος θα αφιερωθεί στην αλλαγή από την έρευνα μέχρι την ε, πρακτική εφαρμογή και την ε, μετάδοση της γνώσης. Έτσι λοιπόν η έρευνα και η καινοτομία θα συνδεθούν πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Πρόεδρε, νομίζω πως για πρώτη παρέμβαση ήταν αρκετά αυτά. Θα χαρώ να απαντήσω στα σχόλια. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα θέμα θεμελιώδου σημασίας και για την αλληλευτική πολιτική. Ήδη στο 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο είχαμε τη δυσάρεστη έκπληξη το τελικό αποτέλεσμα να μην λαμβάνει υπόψη ούτε τα δικά μας αιτήματα και απαιτήσει ούτε καν τις συστάσεις ε, των επιστημόνων που ασχολούνται με εφαρμοσμένη στην αλία έρευνα. Και βλέπω δυστυχώς ότι οι τάσεις αυτές συνεχίζονται, γιατί αυτό που χρειάζεται η αλία είναι σε τελική ανάλυση εφαρμοσμένη έρευνα. Δεν ξέρω, θα το πάρει επιτέλους ποτέ χαμπάρι αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αναφέρεται η αριστεία, η επιστημονική αριστεία ως πρώτος στόχος ε, της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ήδη στο 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο υποχρεωθήκαμε μέσω μιας τροπολογίας στον προϋπολογισμό μέσω σχολείων προσπαθήσαμε να υποχρεώσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική να αφιερώσει ένα ελάχιστο ποσοστό στην εφαρμοσμένη έρευνα για την αλία. Υποτίθεται ότι κόπτεται για την επιστημονική αριστεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού είναι όμως η εφαρμοσμένη έρευνα που είναι η πεμπτουσία και το θεμελιώδη σημείο για την ελευτική πολιτική. Εγώ γνωρίζω προσωπικά πολλούς ερευνητές από ευρωπαϊκά κέντρα, όχι μόνο από ισπανικά, που υπέβαλαν προγράμματα τα οποία απορρίφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώ γιατί τέτοιου είδου εφαρμοσμένη έρευνα δεν εμπίπτει στι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν περιλαμβάνεται. Αυτό για το 7ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο. Ο κύριο Τσουκαλά, που είναι πολύ ε, έμπειρο για τα θέματα αυτά και ε, είχα συνεργαστεί και με τον προηγούμενο εισηγητή για το ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. Ο συντάκτη μα τη γνωμοδότηση έχει πολύ ε, έγκυρες γνώσεις για το θέμα αυτό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και μία βιβλιογραφία και για το 7ο ερευνητικό πλαίσιο που ε, επισημαίνει τα προβλήματα και τις ελλείψεις στην εφαρμοσμένη έρευνα. Ίσως από εκεί θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε κάποιες ιδέες, ώστε επιτέλους ε, να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για εφαρμοσμένη έρευνα στην Αλία. Γιατί για το κεφάλαιο της αλίας ελάχιστα κονδύλια έχουμε για την έρευνα. Ο, η μοναδική πηγή κονδυλίων είναι αυτή. Αν όμως οι επιστήμονές μας, οι ερευνητές μας δεν μπορούν να υποφεληθούν από τα κονδύλια αυτά, προς τι όλες αυτές οι εξαγγελίες. Το να μετράμε τα ψαράκια είναι επιστημονική αριστεία. Το να μετράμε τα ψαράκια για να βρίσκουμε τη βιομάζα είναι επιστημονική αριστεία, ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη και η αρμόδια κατ' ουσίαν Επιτροπή, που δεν είναι δική μας. Αυτά συμβαίνουν και στις ε, πολιτικές έρευνες των κρατών μελών, δυστυχώ. Και εκεί υπάρχει βασικό πρόβλημα έλλειψη εφαρμοσμένη έρευνα. Μην γελά, μην γέλα, μην με κοροϊδεύει. Όχι, με κοροϊδεύει, με κοροϊδεύει. Έχω δίκιο και θέλω να υπερασπίσω τους επιστήμονές μας. Είναι απαραίτητο, γιατί μιλάμε για τα οικοσυστήματα και όλα αυτά, αλλά αν δεν έχουμε χρήματα για την έρευνα που δεν έχουμε, τότε προς τι να τα λέμε όλα αυτά. Έχουμε καταπληκτικούς επιστήμονες, κορυφαίους επιστήμονες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν υπάρχουν κονδύλια για να χρηματοδοτηθεί η έρευνα. Αυτή η κατάσταση κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Θα σα βοηθήσουμε όσο μπορούμε κύριε Τσουκαλά, Σα υποσχόμαστε, σα το υποσχόμαστε, δεν είμαστε πλευρό σα, αλλά πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι για αυτό το θέμα. Κύριε Ντότζ. Ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, θα κάνω μερικά σύντομα σχόλια σε σχέση με αυτά που είπατε. Πιστεύω πως όλοι εδώ συμφωνούμε πως στο μέλλον θα θέλαμε να δούμε μια, έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ελευθερικό τομέα. Η έρευνα και η καινοτομία θα είναι το κλειδί για να το επιτύχουμε αυτό και για να αναπτυχθούν θέσεις εργασίας στον τομέα και στον τομέα της ε, αλλιεύσης και στον τομέα της μεταποίησης. Συμφωνώ με τον συναδελφό μου όσον αφορά τις, με τη συνάδελφο μάλλον όσον αφορά τις ε, δυσκολίες πρόσβασης στο τωρινό πρόγραμμα πλαίσιο 7. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Όταν συνάντησε τους επιστήμονες από τα δικά μας ερευνητικά ιδρύματα στη Βόρεια Ιρλανδία, αυτό έγινε πρόσφατα, ε, αναρωτήκαμε, ψάξαμε να δούμε πώς θα βρούμε χρηματοδότηση για προγράμματα <clears throat> από το πλαίσιο. Και τα προγράμματα αυτά έπρεπε να χρηματοδοτηθούν ε, όπως ε, πρότεινα σε συνεργασία με άλλες χώρες μέσω του προγράμματος πλαισίου. Στο τέλος όμως χρηματοδοτήθηκαν από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ε, εγώ αυτό το θεωρώ αποτυχία. Διότι μπορούσαμε να μάθουμε πολλά εξετάζοντάς το μαζί με άλλα συστήματα διαχείρισης. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό, σε αυτό το σημείο έχει αποτύχει και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το μέλλον, για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Να πω για τον τομέα της ε, μεταποίησης. Ακόμα χρειαζόμαστε έρευνα και καινοτομία. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα του πλαισίου 7. Στη δική μου περιφέρεια, στο δικό μου κράτος μέλος, όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι μικρές και μεσαίες. Και μάλιστα ούτε καν μεσαίες, είναι μόνο μικρές. και δεν μπορούν ούτε να φανταστούν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα πλαίσιο. Θα πρότεινα λοιπόν αυτή εδώ η Επιτροπή πραγματικά να υποστηρίξει τις ιδέες που ανέφερα και η Επιτροπή Γεωργίας και οι άλλες επιτροπές ε, για, τον, για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Ε, το πρόγραμμα πρέπει να απλοποιηθεί, όχι μόνο όμως να απλοποιηθεί επειδή μιλάμε για τις απλοποιήσεις, λες και είναι το ιερό δισκοπότηρο που δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί. Όχι μόνο γι' αυτό. Πρέπει να δοθούν συγκεκρι... Ε, συγκεκριμένες εγγυήσεις για τις ε, μικρές επιχειρήσεις για να έχουν πρόσβαση αυτές στα προγράμματα καινοτομίας και στη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσουκαλάς θέλει το λόγο για να ολοκληρώσουμε. Οι τοποθετήσεις της κυρίας Φράγκα με αναγκάζουν να σας ταλαιπωρήσω δύο-τρία λεπτά για να τοποθετηθώ σχετικά με το γενικό ζήτημα της ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με την έρευνα. Πιστεύω βαθιά ότι η στρατηγική της Λισαβόνας που μολονότι απέτυχε στηρίζεται στη σωστή βάση, δηλαδή στο νέο τρόπο παραγωγής των ανθρώπων, στη βάση της οικονομίας της γνώσης. Στηρίζεται στο τρίγωνο της γνώσης, δηλαδή στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα. Αυτό το τρίγωνο πρακτικός, το οποίο είναι ιδεαλιστικό, στην πράξη είναι ένας μετασχηματισμός χρήματος. Δηλαδή, για να αποκτήσει κανείς γνώσεις μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας, πρέπει χρήμα να μετασχηματιστεί σε γνώση. Από την έρευνα το χρήμα μετασχηματίζεται, η γνώση μετασχηματίζεται σε χρήμα μέσω της καινοτομίας και της καινοτομικότητας. Αυτό είναι το μοντέλο με το οποίο η ανθρωπότητα αρχίζει να παράγει. Πάρα πολύ συχνά γίνεται το σφάλμα να θεωρείτε ότι η καινοτομικότητα συνδέεται αποκλειστικά με τις νέες τεχνολογίες ή τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες όπως φωτονική, όπως βιομηχανική βιοτεχνολογία και ούτω καθεξής όπως επίσης ότι οι ιδέες όπως η αριστεία στηρίζουν μόνο τέτοιου τύπου δραστηριότητες. Θα μου επιτραπεί με αφορμή αυτά που είπε η κυρία Φράγκα να υποστηρίξω και εγώ μαζί της ότι η αριστεία καταρχήν είναι μια ιδιότητα που αναφέρεται σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Είτε κατασκευάζεις παπούτσια, είτε κατασκευάζεις διαστημόπλια, η ίδια αρχή της αριστείας οφείλει να υπάρχει. Στο ζήτημα της Επιτροπής που μας απασχολεί, η θάλασσα στα αλλιεύματα, οι ανθρώπινες ανάγκες, η τροφοδοσία της κοινωνίας αποτελούν σημαντικά ζητήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να παραθεωρούμε. 55 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ετήσιο, ο ετήσιος τζίρος σε αλλιεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εάν μια υδατοκαλλιέργεια πετύχει, και αυτό εξαρτάται από την έρευνα που γίνεται, αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για την ανθρωπότητα, η οποία, να σας θυμίσω, το 2025 θα είναι 8 δισεκατομμύρια και θα έχει μεγάλη έλλειψη κατά κεφαλή θερμίδων ακόμα και για τις αναπτυγμένες χώρες. Άρα οι θάλασσες, τα αλλιεύματα η αηφορία τους, η επιστημονική έρευνα αποτελούν, δεν μπορεί παρά να αποτελούν ένα κύριο σημείο το ίδιο σημαντικό σαν, την, σαν τα φωτοβολταϊκά ή την φωτονική. Αυτές ήταν οι γενικές μου παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε για την κατασκευή μιας έκθεσης που θα υποστηρίζει τις θέσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσουκαλά. Η κυρία Λουβέν ζήτησε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομη. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη για όλο αυτό το σχέδιο για το 2020. Θα ήθελα να ρωτήσω για τη σχέση ανάμεσα στο ΕΤΘΑ και στον ορίζοντα 2020. Ποια είναι η σύνδεση αυτών των δύο. Επίσης θα Ήθελα να πω ότι όχι μόνο η εφαρμοσμένη επιστήμη και η καινοτομία και η ανάπτυξη δεν είναι μόνο αυτοί οι τομείς που ε, έχουμε λήψεις, αλλά και έχουμε λήψεις στους τομείς, στα οικοσυστήματα, στην κλιματική αλλαγή και αυτό πιστεύω κύριε Τσουκαλά θα ήταν χρήσιμο να το τονίσετε στην εκθεσή σας. Ίσως μπορέσουμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Καλώς. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω. Το Συμβούλιο είναι εκεί. Όχι, όχι. Λάθος το ταμπελάκι η Κομισιόν. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα και εγώ να πω λίγα λόγια. Απαντώντας στην κυρία Φράγκα. Ήταν εύστοχα τα σχόλιά της. Όντως υπάρχουν ε, τεράστιες ελλείψεις σε ό,τι αφορά την επιστημονική βάση για τη διαχείριση της αλίας. Αυτό είναι αλήθεια. Αν όμω αναλύσουμε πιο διεξοδικά το θέμα, διαπιστώνουμε ότι αυτέ οι ελλείψει που έχουμε και αυτέ οι αδυναμίε ω προ την επιστημονική βάση ή την έλλειψη επιστημονικών δεδομένων για τη διαχείριση. Υπάρχει, για παράδειγμα, κάθε φορά που οι αρμόδιοι επιστημονικοί οργανισμοί, το διεθνέ Συμβούλιο για την Εκμετάλλευση τη θάλασσα ή η Τεχνική και Επιστημονική Επιτροπή, όταν μα δίνουν έγκυρε γνωμοδοτήσει για τον καθορισμό των τάκ και των ποσοστώσεων ένα μεγάλο υπερβολικό νούμερο. Περίπου το 40% των ηχθιαποθεμάτων για τα οποία προσδιορίζουμε τάκ δεν μπορούν να, αξιολογηθούν η δεδομένων. Υπάρχουν ηχθιαποθέματα για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχουν στοιχεία. Αυτό δεν οφείλεται σε έλλειψη έρευνας υπάρχουν ελλείψεις στο σύστημα συγκέντρωσης των δεδομένων. Αυτό το σύστημα συγκέντρωσης δεδομένων είναι ανεξάρτητο και από το πρόγραμμα πλαίσιο, το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο και από το ορίζοντα 2020. Πρόκειται για άλλο σύστημα που το διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ και επαφίεται στην βούληση των κρατών μελών. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε αυτές τις ελλείψεις στη συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων, θα υποβάλουμε νέα πρόταση για εξυγχρονισμό των συστημάτων και ένα νέο ε, κανονισμό για τη συγκέντρωση δεδομένων που θα είναι πιο αποτελεσματικός, πιο απλός και ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας που μέχρι στιγμής ήταν ο άμεσος συνεργάτης μας για να προσδιορίσουμε τις ερευνητικές προτεραιότητες για ό,τι υπολείπεται από το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά και για το μελλοντικό ορίζοντα 2020 και χάρη στη συνεργασία αυτή νομίζω ότι καθορίσαμε αρκετά εύστοχα τις ερευνητικές μας ανάγκες. Και τονίζω το ερευνητικές. Όχι σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση στοιχείων ή μελετών για την άμεση εφαρμογή του στην διαχείριση ελευτική πολιτική. Γιατί αυτό είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο και όντω υπάρχουν ελλείψει και αδυναμίε. Πάντω, στο θέμα τη έρευνα, Χάρη στην συνεργασία που έχουμε, ε, την αγαστή συνεργασία που έχουμε με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνες... έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα, πολύ χρήσιμο υλικό για την ε, ανάπτυξη των οικοσυστημάτων, για τη διαχείριση ε, ταυτόχρονα πολλών αλληλευτικών ειδών, για τις προστατευμένες θαλάσσιες ζώνες, για την υδατοκαλλιέργεια. Εκεί είχαμε τεράστιες επενδύσεις και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας. Και από αυτή την άποψη, από αυτό το πρίσμα, είναι πραγματικά άμεμπτη η έρευνα που διενεργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο που είναι το σημείο 19 και προβλέπει την τροποποίηση του κανονισμού 1342 του 2008 του Συμβουλίου που προβλέπει μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλληλευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά. Πρόκειται για έκθεση της κυρίας Ντότς. Δεν ξέρω, προτιμάτε πρώτα να λάβετε λόγο η πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πείτε μας εσείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα. Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, συνάδελφοι. Εδώ για το μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλληλευτικές δραστηριότητες ε, που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά, προβλέπουμε την τροποποίηση του κανονισμού βάσει των άρθρων και της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός ε, μας έχει οδηγήσει στο να λάβει μέτρα κατά εξουσιοδότηση και εφαρμοστικά μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Ο κανονισμός της Επιτροπής 2.37-2.10 έχει ληφθεί υπόψη στο πολίτε αυτό το πλαίσιο για τον γάδο. Στα μέτρα του. Όμως το άρθρο 10 του κανονισμού ορίζει ότι εάν υπό το φως των υποστημονικών γνώσεων το ποσοστό θνησιμότητας και τα αποθέματα γόνων δεν είναι πλέον επαρκή, θα πρέπει ο, το Συμβούλιο να αναθεωρήσει τις διαφορές παραμέτρους ώστε το σχέδιο να επιδιώξει τους μέγιστους στόχους του. Ο κανονισμός ισχύει και δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης αυτών των μη καθοριστικών στοιχείων του σχεδίου από το Συμβούλιο. Μια διαδικασία λήψης αποφάσεων βέβαια τέτοια δεν επιτρέπεται βάσει της συνθήκης. Η πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού εκχωρεί τι δυνατότητε αυτέ τροποποίηση ω μη καθοριστικά στοιχεία του κανονισμού, ω μη ουσιαστικά, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τι κατεξοδότηση πράξη μπορεί και άλλε λεπτομέρειε του κανονισμού να αλλάξει, όπω τι τεχνικέ παραμέτρου στο παράρτημα 1, τα παραστεί ανάγκη. Έτσι, προβλέπονται αυστηρέ προποθέσει, μάλλον καλύπτονται αυστηρέ προποθέσει που προβλέπονται ούτω ή άλλω από τον κανονισμό οι κατεξουσιοδότηση αρμοδιότητας θα πρέπει να ανατεθούν και για την προσαρμογή της αλληλευτικής προσπάθειας, ε, καθώς η ομάδα σκαφών μπορεί να μην περιλαμβάνονται στο καθεστώς ε, αλληλευτικής ικανότητας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει την ε, μορφή όπου θα πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες για τα θέματα αυτά και κατά πόσο θα μπορεί να εκχωρεί άδειες ή ειδικέ άδειες πέραν της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που ορίζεται με το άρθρο 30 θα πρέπει όλα αυτά να είναι σαφή μετά τη θέση ίσχυ της συνθήκης της Λισαβόνας. Οι προτινόμενες τροποποιήσεις είναι απαραίτητες αλλαγές που θα επιτρέψουν στο σχέδιο να λειτουργήσει εύρυθμα. Με το νέο πλαίσιο διαδικασία λήψη αποφάσεων, όπω ορίζεται από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Έτσι λοιπόν το σχέδιο τροποποίησης του κανονισμού έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατά πρώτον, χαίρομαι που μας παρουσίασε η Επιτροπή της συλλογιστική της για το θέμα αυτό. Είχα μια σύντομη συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς για το θέμα αυτό. Ελπίζω ότι θα έχουμε και άλλες συνομιλίες όσο προχωράει η διαδικασία. Η Επιτροπή μας είπε πέρα την πρόταση αυτή ως μια απλή μεταφορά του κανονισμού στις διατάξεις με τις οποίες, οι οποίες διέπουν μάλλον τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει τη συνθήκης της Λισαβόνα. Συζήτησα με την Επιτροπή δύο πρώτα σημεία που τα θεωρώ σημαντικά για τη διαχείριση του γάδου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τεχνικό το ζήτημα. Και υπάρχουν στοιχεία με τα οποία μπορώ να συμφωνήσω, άλλα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω. κάποια ευρύτερα μάλιστα ζητήματα γενικότερα που θα πρέπει να τα σχολιάσει ως η Επιτροπή μας σήμερα και άλλα που θα τα δούμε στη συνέχεια της διαδικασίας. Στις 8 Μαρτίου φέτος συναντήθηκαν τα κράτη-μέλη και εκεί υπήρξε συνένεση ότι παρόλο που έχουν προταθεί τεχνικά μέτρα ουσιαστικότερες αλλαγές ε, για το σχέδιο, με το πρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου παραγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει βάσει του άρθρου 34 το όλο σχέδιο να, να προτείνει το 2013, χρόνια μετά την υλοποίηση, την έναρξη υλοποίηση του σχεδίου, δηλαδή ε, κατάλληλε αλλαγέ και προσαρμογέ, παρά τι επιστημονικέ ε, συμβουλέ πέρσι, και παρά την πρωτοπή προ την Επιτροπή από το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Εκεί η Επιτροπή υποσχέθηκε ουσιαστικέ αλλαγές. Η Επιτροπή μας λοιπόν μπορεί να θέλει να το σχολιάσει αυτό, να εκφράσει την άποψή της. Στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Η δεύτερη πτυχή που νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντική και ελπίζω να τοποθετηθεί η Επιτροπή μας, είναι το γεγονός ότι όσο προχωρούμε και γνωρίζουμε ακόμη μια αλλαγή σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, βλέπουμε ότι τελικά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία επί της ουσίας στο Συμβούλιο ή μάλλον μεταξύ Συμβουλίου Επιτροπής και Κοινοβουλίου για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε σε σχέση με τέτοιου είδους σχέδια. Υπάρχουν προγράμματα για το σκουμπρί, για, για το σαβρίδι και για την ρέγκα που θα συμπεριληφθούν στο ίδιο σύστημα. Η Επιτροπή καλό θα ήταν να ερευνήσει και να δει κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια μετακίνηση εδώ καθώς μιλάμε για τα αποθέματα γάδου. Ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων και να συνεργαστώ μαζί τους για να επεξεργαστούμε το ζήτημα. Muchas gracias, señor Señor Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Ντότζ. Όσον αφορά τον σχολιασμό της πρότασης της Κομισιόν, χθε στην ακρόαση συνειδητοποιήσαμε, μας έγινε προφανές πόσο κρίσιμη κατάσταση είναι ο γάδος στην Βόρεια Θάλασσα, δυτικά της Σκοτίας και στην Ιρλανδική Θάλασσα. Και γι' αυτό είναι αναγκαίο, εξακολουθεί να είναι αναγκαίο, να μην γίνουν μόνο αλλαγές στο Ταμείο, αλλά να αλλάξει, να διορθωθεί και το πολιετές πλαίσιο, έτσι ώστε να καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους, τους οποίους μαζί αποφασίσαμε για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Και πιστεύω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας, ότι στην συνθήκη της Λισαβόνας εμείς ως ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή είμαστε πλέον τώρα στη θέση ε, για αυτό το, να λαμβάνουμε πληροφορίες για αυτό το πολιετές σχέδιο από την Κομισιό, να τη συζητούμε και να έχουμε το δικαίωμα συναπόφασης. Ε, με, το Συμβούλιο Λίας ασχολείται τώρα με το άλλο θέμα. Εμείς δεν έχουμε και για το Σολομό δεν έχουμε τόση ε, αρμοδιότητα, όμως εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε και πρέπει να το συζητήσουμε. Και υπάρχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε σημεία που έχουν προταθεί. Ε, δεν θέλω να τα επαναλάβω, αλλά η προσαρμογή των μέτρων είναι αποφασιστικό σημείο, σημαντικό. Ε, η ρύθμιση της, των δαπανών για την αλία επίσης το συζητήσαμε. Συζητήσαμε για την για την ε, χωρητικότητα, για τον ορισμό, για το πόσο σαφής ορισμός πρέπει να είναι, για τον ε, καταμερισμό των δαπανών. Και αυτό επίσης σημαντικό. Αλλαγή των παραρτημάτων. Και πιστεύω πως ορισμένες φορές. Η απόφαση του Συμβουλίου Αλίας βασίζεται σε αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου για, τα, για, για τα αλληλευτικά αποθέματα και αυτό ποικίλει ανάλογα με τα χρόνια. Εγώ μπορώ να πω, για παράδειγμα, είμαι αρμόδιος να μιλήσω για τα ποσοστά στη Βαλτική, για τα αποθέματα στη Βαλτική. Δεν ξέρω όμω τι γίνεται, τι γίνεται στη Βόρεια Θάλασσα. Ξέρω ότι ο γάδο. υπάρχει γίνεται σε... ότι ο γάδο υπεραλλιεύεται στη Βαλτική βρίσκεται, βρίσκεται σε τόσο κρίσιμη κατάσταση που κανονικά θα έπρεπε να απαγορευτεί πλήρω η αλία του, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακάμψει. Τώρα, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε μια αύξηση του γάδου και η Κομισιόν, για να μην, αλλάξει, για να μην αλλάξουν οι τιμές, αποφασίζει να καταστρέψει ορισμένα αποθέματα για να μην πολιθούν και πέσουν οι τιμές. Ε, πρέπει να δείτε, πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, έτσι. Okay. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία. Translation is okay? Yes. Τώρα είναι εντάξει. Συνεχίζω λοιπόν και αυτή είναι η εμπειρία που έχουμε συλλέξει για τον ογάδος. Παρόμοια κατάσταση. Χρειάζεται περιφερειακό σχεδιασμός και περιφερειακή διαχείριση. Εκεί πολιεύονται αυτά τα ψάρια όχι αλλού, όχι κεντρικά. Ο Γάλλος συνάδελφος ε, μας μίλησε για το τρίγωνο Ιρλανδία, Σκοτία, Αρκτικός, Αρκτικός ωκεανός. Μας είπε τι γίνεται εκεί, ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται ώστε να ανακάμψει κάπως ο πληθυσμός και φυσικά όλα αυτά παίζουν ρόλο. Μιλάτε για πράξεις κατά εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως μην ξεχνάμε, πρέπει να, πετήσουμε, να πετούμε κάθε χρόνο μία έκθεση για, τα, για τον πληθυσμό του γάδου σε αυτές τις περιφέρειες ε, και σε αυτές τις περιοχές αλίας. Μόνο έτσι θα γίνει η δουλειά. Ευχαριστούμε κύριε Κούν, κύριε Λοβέν. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ και την κυρία Ντότζ που έθεσε το θέμα επιτάπητος. Ε, αν κατάλαβα καλά, η πρόταση είναι να ευθυγραμμιστεί αυτό το σχέδιο διαχείρισης με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό που διακυβεύεται λοιπόν εδώ είναι το αν εμείς συμφωνούμε με τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις και τις ε, εκτελεστικές πράξεις και είναι πολύ βασικό θέμα για αυτήν εδώ την Επιτροπή. Διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μέση αυτού του παιχνιδιού εξουσίας με τα όργανα. Δεν ήμουν εισηγήτρια σε κανένα από αυτά τα... σε καμία από αυτές τις εκθέσεις, οπότε δεν είμαι νήμερη για όλες τις ε, λεπτομέρειες, αλλά πιστεύοντας την κυρία Ντότς και στην άποψή της ε, για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Πιστεύω ότι οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση μπορούν να ανασταλούν από το Κοινοβούλιο. Δεν εξουσιοδοτούμε μέσα την Κομισιόν. Αν θέλουμε να, σταματή, να τη σταματήσουμε, τη σταματάμε. Εγώ δεν βλέπω κάτι επικίνδυνο στην, ε, στις πράξεις κατά εξουσιοδότηση στην Κομισιόν τώρα όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις. Και η εναρμόνιση των μέτρων για να είναι τα ίδια για όλα τα κράτη-μέλη. Σε μένα φαίνεται λογικό οι αλληλευτικές άδειες και η ανταλλαγή πληροφοριών να εναρμονιστούν. Πραγματικά όμως θα ήθελα να μάθω τι πιστεύει και η κυρία Ντότζ για αυτό. Γενικά πάντως να επιστήσω την προσοχή. Χρειαζόμαστε να είμαστε προσεκτικοί και με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή για τα ζητήματα αυτά. Διαφορετικά δεν θα έχουμε κανένα σχέδιο διαχείρισης ούτε τώρα ούτε μετά τη μεταρρύθμιση της, ε, της ΚΑΛΠ. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε κύριε Λεβέν. Θέλει το λόγο κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι η κυρία Ντότς. Θέλετε κυρία Ντότς να δευτερολογήσετε, ναι. Να επανέλθω σε αυτά που είπε η Ζαμπέλ. Εξετάσαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και κατά τη γνώμη μου, αν συμφωνήσουμε σε ένα σχέδιο, και νομίζω ότι όλοι εδώ στην Επιτροπή συμφωνούμε ότι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης είναι η κατάλληλη λύση. Γιατί η, ε, η τωρινή πρακτική με αλλαγή κάθε και παζαρέματα κάθε Δεκέμβριο είναι εμφανώς ακατάλληλη. Οι επιχειρήσεις και οι λύσεις δεν μπορούν να κάνουν μια πιο μακροπρόθεσμη οργάνωση και ένα μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης που θα έχει ε, αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συντονισμού. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Ένα τέτοιο μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης που θα το έχουν διαπραγματευτεί Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, συνεργασία, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας δώσει καλύτερη ε, άποψη για το πως θα που η αλληλεία. Τώρα, για το κατά πόσο θα έχουμε κατεξουσιοδοί εφαρμοστικέ πράξει. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, εξαρτάται από το τι πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για το σχέδιο. Κάποια στοιχεία του σχεδίου έχουν πιο μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα, ίσως χρήζουν, χρήζουν κάποιες προσαρμογής. Αλλά δεν είναι θεμελιώδη σημασία για τη γενική πορεία του σχεδίου. Νομίζω ότι έτσι αποσαφηνίζεται η προσέγγιση μας για το ποια άγουσα θέλουμε να ακολουθήσουμε. Καλώς, πάμε στο επόμενο σημείο, το 20. Το πολιετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική και τις αλλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύεται από θέματα αυτατροπής του κανονισμού 1098 του 2007. Ε, ρώτησα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είδα αντίδραση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τα σχόλιά της και να διευκρινίσω ότι η πρόταση αυτή είναι μία από την πληθώρα προτάσεων που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλουμε μία ευθυγράμμιση, γενική ευθυγράμμιση της ε, νομοθεσίας μετά τις ε, κατευθυντήριες γραμμές της συνθήκης της Λισαβόνας. Και αυτή η πρόταση ακριβώς δίνει μια απάντηση στο θέμα της ευθυγράμμισης. Έχει απόλυτο δίκιο η συγγετρία ότι υπάρχει ένα άλλο όμιζο πρόβλημα με τη μακροπρόθεσμη διαχείριση και το μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης ε, γάδου στη Βόρειο Θάλασσα και σε άλλες περιοχές. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, του ενδιαφερόμενους, τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια και την Επιστημονική Επιτροπή, προκειμένου να αναζητήσουμε την πιο κατάλληλη λύση για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα αυτού του μακροπρόθεσμου σχεδίου διαχείρισης. Ήδη έχει γίνει μια αξιολόγηση του σχεδίου και στην αξιολόγηση αυτή εντοπίστηκαν πολλά νευραλγικά σημεία για την βελτίωση του σχεδίου. Επίσης, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους στα κράτη-μέλη, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μία σωστή λύση θα ήταν να προετοιμάσουμε ένα μεικτό σχέδιο αλίας, γιατί ένα μείζον ζήτημα είναι οι Επειδή η κατάσταση στην αλία είναι μεικτή, δεν αλλιεύεται ποτέ ένα, μόνο αλλιευτικό είδος. Οπότε μακροπρόθεσμα θα πρέπει να εντοπίσουμε ένα σχέδιο μικτής αλίας. Και η Επιστημονική Επιτροπή επεξεργάζεται αυτό το θέμα, θα υποβάλει συστάσεις και με βάση αυτή τη γνωμοδότηση θα υποβάλουμε και εμείς πρόταση. Πάντως θα συνεχιστούν οι συζητήσεις με το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και τους ενδιαφερόμενους για το ποια θα πρέπει να είναι τα κεντρικά σημεία αυτού του νέου σχεδίου. Βέβαια, η Επιστημονική Επιτροπή θέλει κάποιο χρόνο για να προτείνει κάποιες τεχνικές λύσεις. Και ίσως ε, η Επιτροπή, μετά από έτσι των κρατών μελών, θα υποβάλει ε, εντό ολίγου μια μικρή εμβέλειας ε, αναθεώρηση με διευκρινήσεις για κάποια άρθρα και επεξηγήσει για το θέμα της ελευτική προσπάθειας. είναι όμω περιορισμένη εμβέλεια αυτή η πρόταση, γιατί πιστεύω ότι για να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα του σχεδίου θα πρέπει στο μέλλον να έχουμε ένα τέτοιο σχέδιο διαχείρισης ε, που να αναφέρεται σε μεικτή αλλιεύση. Επίσης, στην πρότασή μας θα πλουστεύσουμε και θα εξηγήσουμε και κάποια άρθρα. Πάντως, το μείζον πρόβλημα της συγκεκριμένη πρότασης αφορά την ευθυγράμμιση με τη νέα συνθήκη, τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πάντως, ε, θα επανέλθουμε και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο με νέες προτάσεις για ένα πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης. Ευχαριστώ. Ωραία, τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 20 το πολιετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική και τις αλλιευτικές δραστηριότητες ε, εκμετάλλευση αυτών των αποθεμάτων. Ε, η συγκεκριτής είναι ο κύριος Βαγουένσα. Θα ακούσουμε όμως πρώτα την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Βαγουένσα και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε, δεν χρειάζεται καν να επαναλάβω αυτά που είπα και προηγουμένως για το σχέδιο διαχείρισης για τα αποθέματα γάδου στη Βόρεια Θάλασσα. Το ίδιο ισχύει και για τη Βαλτική. Πρόκειται για μία πρόταση ευθυγράμμισης. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας έγινε αξιολόγηση του σχεδίου αυτού και μετά από επανειλημμένα αιτήματα των κρατών μελών και του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική επεξεργαζόμαστε ένα νέο σχέδιο. Στο μεταξύ όμω. και σύμφωνα με το αίτημα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου υποβάλαμε αυτή την πρόταση προκειμένου να αλλάξει η διαδικασία λήψη αποφάσεων. Προς το παρόν δεν έχω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαγουένς έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φάνηκε και από το προηγούμενο σημείο ότι ενώ αρχικά είχαμε ε, μόνο ένα θέμα ευθυγράμμισης με τη συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να πάει λίγο πιο μακριά και προ... το... πρότεινε και τροποποίηση του κανονισμού και των προθεσμιών ε, αξιολόγησης. Δεν ξέρω αν έχει νόημα, στα πλαίσια αυτή τη ευθυγράμμιση, να ασχοληθούμε και κάποια προβληματικά σημεία του κανονισμού και να προτείνουμε και άλλε τροποποιήσει, γιατί ο κανονισμό είναι παροχημένο και δεν ανταποκρίνεται στην παρούσα κατάσταση τη βαλτική. Ούτε λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων αλληλευτικών ειδών. Γιατί το πολιτές ε, σχέδιο για τα αποθέματα γάδου μερικές φορές ε, ε, οδήγησε στην, στον περιορισμό των αποθεμάτων, γιατί δεν υπάρχει ελαστικότητα, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε τα επιστημονικά πορίσματα, είτε οι απόψει των ε, αλλιών που λένε ότι η κατάσταση αποθεμάτων βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ω προ το γάδο. Και από αυτήν την άποψη οι αλλιευτικέ ποσοστώσεις μπορούν να αυξηθούν και κατά 40%. Με βάση όμως αυτό που προβλέπει το πολιτικό σχέδιο που εκ των προτέρων ε, προσδιορίζει τις ελευτικές ποσοστώσεις και τον μπλοκάρει σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται με την πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε αύξηση των ποσοστώσεων πέραν του 15 προβλεπόμενου τα 100. Οπότε έχουμε την εξή κατάσταση. Τα αποθέματα του γάδου βρίσκονται σε καλή κατάσταση στη Βαλτική, κάτι που είναι καλό για την αλίευση, αλλά υπάρχει πρόβλημα με την ύπαρξη της, ε, με την επιβίωση των αποθεμάτων σαρδελόρεγγας αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ληφθεί υπόψη και να προβλεφθεί μια μεγαλύτερη ελαστικότητα σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των ΤΑΚ. Γιατί με βάση τα επιστημονικά πορίσματα, τα εκθεαποθέματα γάδου ε, ε, τηρούν τα, τις απαιτήσεις της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και η θνησιμότητα που είναι χαμηλή μας επιτρέπει να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τα τάκ για το γάδο πάνω από 15%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ε, δεν ε, υπέβαλε την πρόταση που είχε υποσχεθεί για την ε, μεγαλύτερη ελαστικότητα του πολίτου σχεδίου. Θα πρέπει να αυξηθεί η ποσόστοση πάνω από 15% εφόσον το από γάδο το επιτρέπει. Και ε, Ακριβώς ε, επειδή πελαγικά είδη που έχουν αλληλεπίδραση με το γάδο μειώνονται στο μέτρο που ο γάδος, τα αποθέματα γάδου αυξάνονται. Γι' αυτό θα πρέπει να λιεύεται πολύ περισσότερο. Επίση, ε, έγινε μια παράταση από 3 σε 5 χρόνια για την εξέταση. Είναι υπερβολικά μακροπρόθεσμη αυτή η προθεσμία για την ε, προσαρμογή του σχεδίου στις εξελίξεις ε, της κατάστασης στη Βαλτική που είναι πολύ δυναμικές. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτή την παράταση από 3 σε 5 χρόνια. Δεν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ένα πολιτές σχέδιο δεν θα πρέπει να είναι κάτι άκαμπτο, ιερό και απαράβατο, αλλά να γίνει ένας ε, μηχανισμός ελαστικός που θα μπορεί να επιτρέπει την προσαρμογή των αλληλευτικών προσπαθειών ε, στα επιστημονικά πορίσματα και την επιστημονική γνώση. Αυτά. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε πολύ ψωμί να φάμε με αυτή τη γνωμοδότηση. Ευελπιστώ πάντως ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ιδιαίτερα για τα πιο φλέγοντα ζητήματα αυτού του θέματος. Ευχαριστούμε κύριε Βαγουέσα, η κυρία Λόβιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να λάβω το λόγο αυτή τη στιγμή, διότι ε, πίστευα πως θα μιλούσαμε μόνο για την εναρμόνιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά τώρα μεταράξατε. Αναστατώσατε. Λοιπόν, μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης. Αυτό το σχέδιο ε, έχει γίνει έτσι ώστε η... ο αλληλευτικός τομέας να μπορεί να σχεδιάσει μακροπρόθεσμα. Μέχρι τώρα η διαχείριση δεν επέτρεπε στην αλληλευτική βιομηχανία να σχεδιάζει οικονομικά μακροπρόθεσμα. Δεν μπορούσε να ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Οι ποσοστώσει αυξήθηκαν κατά 100% ε, ένα χρόνο, μετά τον επόμενο μειώθηκαν κατά 80% και αυτό είχε καταστρέψει τη βιομηχανία. Δεν ήταν καλό. Το μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης τώρα στη Βαλτική αυξάνει τα ηχθιαποθέματα γάδου προς όφελος της ε, βιομηχανίας αλίας γάδου, προς το μελλοντικό της όφελος. Όλοι ξέρουμε εδώ πως ο γάδος μπορεί να φτάσει τα 50 χρόνια ζωής. Θέλουμε να υπάρχουν αυτά τα μεγάλα ψάρια για να μπορούν να αναπαραχθούν στη Βαλτική, έτσι ώστε να αυξηθεί ο πληθυσμός του γάδου στη Βαλτική. Και ανησυχώ με αυτά που λέτε εδώ ότι ο γάδος τρώει τη σαρδελόρεγγα και κινδυνεύουν έτσι οι μεγάλες μηχανότρατες που ψαρεύουν σαρδελόρεγγα. Έχουμε μια πολιτική επιλογή να κάνουμε εδώ πέρα. Θέλουμε να προωθήσουμε τον γάδο που, προτίθε, που ε, προ, ε, προορίζεται για κατανάλωση ή θέλουμε να προωθήσουμε τις μηχανότρατες που ψαρεύουν για να ταΐσουν τους σολομούς στις νορβηγικές υδατοκαλλιέργειες. Υπάρχει στη Βαλτική μια προφανής διαμάχη συμφερόντων. Όταν... Και είναι προφανές επίσης ότι αν μειωθεί ο γάδος θα υπάρχει περισσότερη σαρδελόρεγγα. Δυστυχώς, αυτό που κάναμε με το να εξαντλήσουμε σχεδόν τα αποθέματα του γάδου είναι να επενδύσουμε σε άλλα αλευτικά σκάφη τα οποία θέλουν να συνεχίσουν να ψαρεύουν της Αρδελόρεγκα. Αλλά θα προτιμούσαμε να, υπάρχει, να υπάρχουν υγιείς γάδοι στη Βαλτική, όπως ήταν κάποτε τη δεκαετία του 80, αντί να έχουμε ξένο σολομό που έχει τραφεί με δικές μας αρδελόρεγγες. Ε, σας παρακαλώ να το συζητήσουμε αυτό ήρεμα. Ε, πιστεύω ότι η εναρμόνιση του ισχύοντος σχέδιου για το γάδο είναι θέμα μιας άλλης συζήτηση την οποία πρέπει να διεξάγουμε με λεπτομέρειες δημόσια. sorry for... Λυπάμαι για την... που μακρηγόρησα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Yes. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μερικές σκέψεις για αυτά που ακούσαμε. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Ναι, πράγματι τροποποιήσαμε το στόχο του σχεδίου. Πράγματι εισαγάγαμε το στόχο της, ε, του να ψαρεύουμε τα αποθέματα γάδου. Ένα από αυτά τα αποθέματα έχει διφτάσει στο όριο που μπορούμε να αλλιεύσουμε και δυστυχώς πράγματι παραδέχομαι ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση ή μείωση στις ε, ποσοστώσεις κάθε χρόνο. Κατά 15% και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τον αληφτικό τομέα να σχεδιάζει από πολύ νωρίτερα τις δραστηριότητε του. Σήμερα θα δημοσιευτεί μια επιστημονική σύσταση για τη φετινή χρονιά Δυστυχώ όμως δεν θα είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα για το γάδο όπως ήταν πέρυσι. Αλλά είναι προτέρημα να έχουμε μακροπρόθεσμο σχέδιο για να μην απομακρυνθούμε πολύ από το όριο του 15% στις αυξομοιώσεις για το γάδο. Το πρόβλημα με το μακροπρόθεσμο σχέδιο και την καρτάρτισή του που διαπιστώσαμε πρόσφατα είναι ότι εάν τεθεί μια προθεσμία για αξιολόγηση, για παράδειγμα, σε δύο χρόνια από τώρα, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε το σχέδιο αντικειμενικά και δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις στα, στα ηχθή του γάδου. Μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε τις επιστημονικές εκθέσεις που έγιναν γι' αυτό και θα δείτε ότι τα δύο χρόνια είναι πολύ μικροχρονικό διάστημα για να αξιολογήσουμε σωστά τα μέτρα. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι το ε, μακροπρόθεσμο σχέδιο είχε κάποια επιρροή στα εχθή αποθέματα. Είναι καθήκον της ISIS, της υπηρεσίας αυτής, να παρατηρεί, να ελέγχει το καθεστώς των αποθεμάτων στη θάλασσα και να δημοσιεύει επιστημονικές συμβουλές και επικαιροποιημένε επιστημονικές εκθέσεις. Υπάρχουν ρήτρες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπου εμείς μπορούμε να επέμβουμε νομοθετικά εάν προκύψουν απροσδόκητες αλλαγές. Και, τελευταίο σχόλιο, Πράγματι, εμείς εργαζόμαστε πάνω σε ένα νέο σχέδιο, το οποίο θα λάβει υπόψη όλες τις διαδράσεις ανάμεσα στα είδη των ψαριών, όπως είπατε πριν. Στην τελευταία έκθεση μπορούμε να διαβάσουμε ότι υπάρχει μία ανάγκη για πρόσθετες επιστημονικές πληροφορίες. και καθώς επίσης ότι υπάρχει μια ανάγκη για συζητήσεις, για διαβουλεύσεις με το κοινό, οι οποίες δεν έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα. Όμως τώρα είμαστε ακόμα στο πρώτο στάδιο. Θα προχωρήσουμε και ελπίζουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη να φτάσουμε σε ένα νέο σχέδιο. Ευχαριστούμε κύριε Βαγουένσα. Έχετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, τέλεια. Οπότε ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο, το σημείο 15 δηλαδή τη ημερήσια διάταξη. Το πολιτέ σχέδιο για το απόθεμα Σολομού τη Βαλτική και την αλίευση του συγκεκριμένου εχθή αποθέματο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου μας παρουσίασε την πρότασή της και σήμερα θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Γκρουμπάρτζικ, που θα μας παρουσιάσει την έκθεση του. Έχετε το λόγο κύριε Γκρουμπάρτζικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του γάδου, αλλά είναι τόσο ευρύ το ζήτημα αυτό και θα έχουμε χρόνο να επανέλθουμε στο ζήτημα άλλη φορά. Οπότε ας περιοριστούμε στο σολομό της Βαλτικής αυτή τη φορά. Σας ε, υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες συμβιβαστικές μετά από τις τροπολογίες ε, που κατατέθηκαν και τις αντιδράσεις μας ε, ως προς την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έγινε και ανταλλαγή απόψεων με τους και ηγητές και έγινε και συζήτηση από την οποία προέκυψαν πολύ βασικά σημεία για το πολιετές σχέδιο προστασίας του Σολομού της Βαλτικής, ε, γιατί ε, διαφωνούμε ε, με τις αδερές γραμμές πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλουμε να τροποποιήσουμε την πρότασή της. Η διαβούλευση ήταν ευρεία και επαναλαμβάνω ότι το Περιφερειακό Συμβουλευτικό Συμβούλιο για τη Βαλτική είχε ριζικά αντίθετη άποψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αντίθετη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλευτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική δείχνει ότι ο αλληλευτικός κλάδος και όχι μόνο αυτό γιατί το ΡΑΚ έχει ευρύτερε αρμοδιότητες σημαίνει ότι ε, διαφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έδειξαν και οι διαβουλεύσεις. Ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γνώμη του κλάδου και του Περιφερειακού Συμβουλευτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική Θάλασσα και η αισθητή διαφωνία. Φαίνεται όμω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδιαφορεί πλήρω για τη θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου, του ΡΑΚ. Κάτι που δεν συνάδει με την κοινή αλληλευτική πολιτική και με την ε, πρόταση για την περιφερειοποίησή τη. Οι τροπολογίε μα αφορούν ε, διάφορα σημεία τη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καταρχήν είχαμε την πρόταση της Επιτροπής που αφορούσε τον ε, εμπλουτισμό και τον καθορισμό, τον ορισμό των ε, ποταμών πλούσιων σε Σολομό. Ε, προτάθηκε μετά από μία επταετία να σταματήσει, να διακοπεί η διαδικασία του εμπλουτισμού των αποθεμάτων και μάλιστα χωρίς όρους. Εκ των προτέρων προσδιορίστηκε ε, ο αριθμός και οι τοποθεσίες ε, ποταμών πλούσιων σε ε, Σολομό, σε άγριο Σολομό, προτάθηκε η επταετία και αποκλείστηκαν άλλοι ποταμοί. Αυθαίρετα όμως. Σε ό,τι αφορά το σημείο, το άρθρο 14, υπάρχει ένα μεταφραστικό λάθος. Εκεί αναφέρεται ότι ο εμπλουτισμός ε, θα εξαρτηθεί από το επίπεδο παραγωγής. Αν το επίπεδο παραγωγής ε, σε συγκεκριμένο ποταμό δεν φτάνει στο 80% της δυνητικής παραγωγικής ικανότητας, τότε θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία του επανεμπλουτισμού. Γιατί στόχος μας είναι στα... να υπάρχουν πολύ περισσότεροι ποταμοί πλούσιοι σε Σολομό, πολύ περισσότεροι από ό,τι υπάρχουν σήμερα γιατί από ιστορική άποψη η Βόρεια Ευρώπη ήταν γεμάτη από ποτάμια πλούσια σε σολομούς. Γιατί να περιορίσουμε τον αριθμό των ποταμών αυτών και μάλιστα αυθαίρετα. Δεν, δεν συνάδει αυτό με την πρόθεση των χωρών μελών, γιατί νομίζω ότι έχουν συμφέρον τα κρατη να έχουν ποτάμια που θα είναι γεμάτα, θα βρίθουν σολομού. Επίσης, ε, προτείνω δεκαετία για, την, για τον επανεπλουτισμό σε περίπτωση που ε, επιτευχθεί το 80%. Αν δεν επιτευχθεί όμως, να γίνουν μελέτες από τις χώρες ε, που να δείχνουν γιατί δεν έχει υλοποιηθεί το ποσοστό το 80%. Και θα πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Γιατί δεν γίνεται επανεμπλουτισμός ε, σε ποτάμια που είναι ακατάλληλα για αναπαραγωγή και μάλιστα έγιναν ε, έρευνες από επιστήμονες και κάθε χώρα γνωρίζει ποια ποτάμια της ε, προσφέρονται για την αναπαραγωγή του σολομού. Μετά την άρση των εμποδίων που μπλοκάρουν τον επανεμπλατισμό σε αποθέματα, θα πρέπει να περιμένουμε μία ακόμη δεκαετία για να υλοποιήσουμε το συντελεστή του 80%. Και μετά την υλοποίηση αυτού του συντελεστή του 80%, θα έχουμε επιτέλους ένα ποταμό που θα είναι πλούσιος σε σολαμό και διακόπτεται η διαδικασία του επανεμπλωτισμού εφόσον ε, η χώρα, η Κομισιόν αναγνωρίσει ότι αυτός ο ποταμός είναι πλέον ε, πλούσιος σε σολομό. Αλλά το κράτος θα πρέπει να έχει την υποχρέωση να μεριμνά ώστε να διατηρηθεί αυτή η αυθονία του σολομού στο συγκεκριμένο ποταμό. Άλλο σημείο αφορά κάτι που συζητήσαμε και προηγουμένως, την αλία μικρής κλίμακας ή την ερασιτεχνική αλία και την ε, υποχρέωση τήρηση ημερολογίων πλοίου ε, προαναγγελίας. Εδώ προτείνω ε, να λάβουμε υπόψη τα πλοία άνω των 12 μέτρων, όπως προβλέπει ε, η μικρή κλίμακα σαλία. Τα λευτικά σκάφη μήκο μικρότερο των 12 μέτρων θεωρούνται ω ε, λευτικά σκάφη μικρή κλίμακα αλεία και άρα δεν υπόκεινται στην υποχρέωση τη στήριξη ημερολογίου γιατί ασχολούνται κυρίω με την παράκτια αλία. Ένα άλλο θέμα είναι η ερασιτεχνική αλία. Η αριστεχνική αλία και η αλήψη Σολομού σε αυτά τα πλαίσια είναι προβληματική. Και μάλιστα από τη χθεσινή δημόσια κρόαση διαπιστώσαμε ότι στην ε, Ιταλία είναι εύκολο να κανεί αριστέχνη γιατί δεν χρειάζεται να το δηλώσει και αποφεύγει και του ελέγχου. Είναι τελείω ανεξέλεγκτη η αριστεχνική ελία, οπότε συμφέρει κανεί να είναι αριστέχνη αλληλή παρά να δηλώνει ότι είναι επαγγελματία ε, ψαρά. Γιατί όταν είναι επαγγελματία κανεί ο ψαρά, υπόκειται σε δρακόντιου και πολύ τακτικού ελέγχου. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε πώ θα αντιμετωπίσουμε την άρεση τεχνική και να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση τη αερασιτεχνική αλεία. Ώστε όσοι αλλιεύουν αερασιτεχνικά για λόγους αναψυχής να ελέγχονται επίσης εφόσον αλλιεύουν σολομούς για να μην καταλήξουμε σε παράλογα αποτελέσματα ώστε κάποιος που θέλει με καλάμι να ε, αλλιεύσει να χρειάζεται ειδική αλλιευτική άδεια. Ήδη έχουμε τον κανονισμό 1224 του 2009 και το 404 του 2011. Οι δύο αυτοί κανονισμοί προσδιορίζουν τον τρόπο χορήγησης των αδειών σε περίπτωση αεραστεχνικής αλίας ή αλίας για λόγους αναψυχής και σας παραπέμπω σε αυτούς τους δύο κανονισμούς. Τώρα, το θέμα της νομιμότητας και την ανάγκληση της εξουσιοδότησης, της κατεξουσιοδότησης πράξης ή τα τεχνικά μέσα που προσδιορίζονται από τα κράτη-μέλη θα ελέγχονται όχι στη διάρκεια της τριετίας αλλά μέσα σε ένα χρόνο. Κάτι που είναι λογικό για να μπορούμε να αντιδρούμε εγκαίρως στις αλλαγές. Νομίζω ότι απαιτείται μια τέτοια ελαστικότητα, γιατί είναι δυναμική η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώς ε, με πολύ περίπλοκο τρόπο ε, ελέγχει την ε, νομιμότητα. Αρχικά ήταν έξι χρόνια, τώρα αναφέρονται τρία δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό το θέμα, αυτή η σωστή προσέγγιση. Το θέμα της ανάκλησης εξουσιοδότησης ε, ήταν ιδιαίτερα επίμαχο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών να μπορεί να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση. Θα πρέπει σε τέτοια περίπτωση να ανατρέξουμε στη συνθήκη της Λισαβόνας και να εφαρμόσουμε εκείνη τη διαδικασία ως προς την ανάκληση της εξουσιοδότησης που χορηγείται στα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι η δεσμευτική νομοθεσία. Και το τελευταίο θέμα είναι οι θηρευτές, οι φυσικοί εχθροί των αποθεμάτων Σόλωμου της Βαλτικής. Ξέρω ότι διαφωνούμε με την Ισαβέλα Λαβίν και εγώ είμαι ε, θερμός υπέρμαχος ε, της φώκιας, αλλά έχει αποδειχθεί από όλες τις ε, επιστημονικές μελέτες που εξέτασα, καταλήγουν δεν, δίνουν, δεν αντανακλούν την πραγματικότητα της Βαλτικής. Αναφέρεται ότι η επιρροή των φωκιών και των κορμοράνων, βέβαια με τους κορμοράνους ισχύει τελείως διαφορετικό θέμα, αλλά ε, και η φωκή είναι προστατευμένο είδος και δεν αναφέρεται σε επιστημονικές μελέτες ποια ακριβώς είναι η επιρροή τους στα αποθέματα Σολομού. Πιστεύω ότι και αυτές θα πρέπει να αναφερθούν, να περιληφθούν στην πρόταση για την αξιολόγηση των αποθεμάτων. Και μετά από τρία χρόνια θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την επίδραση των φυσικών εχθρών, των θηρευτών, ιδιαίτερα των φωκιών και των κορμοράνων, για να δούμε πώς επηρεάζουν τα αποθέματα Σολομού. Και μέχρι το 2016 να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο διαχείρισης. Αν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους θηρευτές αυτούς, τις φώκες και τους κορμοράνους, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα υπερασπίσω τα δικαιώματά τους και θα ταχθώ υπέρ αποφυγής οποιασδήποτε επέμβασης στο οικοσύστημα. Ευχαριστώ κύριος Βαγουένσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Γκρουμπάρτζη και την πολύ καλή του έκθεση. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό θέμα είναι το θέμα του επανεμπλωτισμού των αποθεμάτων αναφέρθηκαν κάποια πολύ αρνητικά σχόλια για τον επανεμπλουτισμό. Δεν συμφωνώ ότι θα πρέπει να απαγορεύεται ο επανεμπλουτισμός 7 χρόνια μετά τη θέση ισχύ του κανονισμού. Οι διατάξεις που τίνουν σε κατάργηση του επανεμπλουτισμού ε, ε, νομίζω ότι δεν θα είναι αποτελεσματικές γιατί είναι πραγματικά πολύ ε, μεγάλη ανθρωπογενή επιρροή στα αποθέματα του Σολομού. Επίσης, ε, θα πρέπει να αναζητήσουμε καλύτερη ποιότητα ε, του γενετικού υλικού του επανεπλατισμού και να καταργήσουμε τις, τον ακατάλληλο επανεπλουτισμό. Γιατί ένας ακατάλληλος επανεπλουτισμός μπορεί να έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα για την βιοπικιλότητα στα οικοσυστήματα όπου υπάρχουν και σολομοί. Και σε περίπτωση ε, τέτοιου ανακατάλληλου αναπληκτισμού θα οδηγόμαστε σε εξαφάνιση του σολαμού σε πολλά ποτάμια. Και μάλιστα οι προτάσεις ε, του κανονισμού για, που αναφέρονται ε, σε επανεπλουτισμό μόνο σε πλούσιους σε σολομό ποταμούς ή τις ενδιάμεσους επανεπλουτισμούς για δυνητικά πλούσιους σε σολομό ποταμούς. Θα ήθελα να πω ότι οι προτινόμενοι περιορισμοί οδηγούσαν στο αποτέλεσμα ε, να έχουμε επιρροή στις ε, αποδημητικές τάσεις των ε, κοπαδιών του Σολομού. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις επιστημονικές μελέτες ό,τι αφορά την αποκατάσταση των αποθεμάτων Σολομού, ιδιαίτερα σε ποτάμια που υπάρχει ιστορική παρουσία Σολομού, γιατί πολλές φορές εξαιτία της ανθρώπινης επιρροής είχαμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Ε, δυστυχώς ε, αν εξαφανιστεί σολομός από τα μένα αυτά θα πληγούν η φύση, το περιβάλλον, ε, η τουριστική ελεία αναψυχής και φυσικά και οι ψαράδες που αλλιεύουν σολομούς. Θα πρέπει να μην συνεχιστούν οι αρνητικές επιδράσεις στο οικοσύστημα και στους τόπους αναπαραγωγής σολομών. Είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Ούτε συμφωνώ με την πρόταση για αυστηρότερου ελέγχου των αλλιευμάτων, τουλάχιστον το 50% των εκφορτώσεων. Το, ο κανονισμό 1224 του 2009, που μιλάει για το ενιαίο σύστημα ελέγχου για τη διαχείριση της αλληλευτικής πολιτικής, περιλαμβάνει άλλο ποσοστό που είναι καλύτερο. Ε, το ίδιο ισχύει και το άρθρο 17, που μιλάει για τους ελέγχους. Με βάση την πρόταση, οι κυβερνήτες ελευτικών σκαφών θα πρέπει να δηλώνουν τα ελεύματα αμέσω μετά την ολοκλήρωση ελευτικής προσπάθειας. Αυτό είναι ουτοπιστική διάταξη. Θα πρέπει να τροποποιηθεί αυτή η διάταξη. Επίσης, ε, διαφοροποίηση βιομηχανικής και αεραστεχνικής αλίας. Χαίρομαι που προτείνει σημαντικές διατάξεις για την αεροσιτεχνική αλεία. Επίσης, ε, συμφωνώ με τα σχόλιά του σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της χρήσης παρασυρώμενων δικτυών και το θέμα του διακαίνου που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Μία παρατήρηση τώρα όχι προς τον εισηγητή μας, αλλά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι πλήρης ο κανονισμός και να εξυπηρετήσει πραγματικά και το περιβάλλον και τους αλείς, θα πρέπει να αλλάξει τελείως ε, ε, πρίσμα αυτός ο κανονισμός, για να μην πω ότι θα πρέπει να αναδιατυπωθεί. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις ο κανονισμός είναι μη ρεαλιστικός. Γιατί δηληθήκε υπόψη ο κανονισμός 11.00 ε, που αναφέρεται στην ανασύσταση των αποθεμάτων ε, χελιού. Είναι πολύ πιο δόκιμες εκείνες οι διατάξεις παρά η διατάξη του τελευταίου κανονισμού που είναι υπερβολικά περίπλοκος και άσχετος με την πραγματικότητα. Θα ήθελα να πω ότι περιμέναμε εδώ και καιρό τον κανονισμό αυτό, αλλά δυστυχώς μας απογοήτευσε τα μάλα. Αν εγκριθεί με τη μορφή που έχει, θα έχει πολύ αρνητικό αποτέλεσμα και στα ηχθιαποθέματα Σολομού και στις αλληλευτικές κοινότητες. Ευχαριστούμε κύριε Βαγόνισσα, ο κύριος Κρίστανσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή για τη δουλειά του στο θέμα της έκθεσης αυτής. Και εγώ ανησυχώ με την έλλειψη επιστημονικών δεδομένων σε αυτόν τον τομέα. Στην ακρόαση βεβαίως ακούσαμε τους ε, εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο προετοιμασίας αυτού του, αυτής της έκθεσης. Ο συνάδελφος εδώ βρήκε κάπως ε, σοβαρές πληροφορίες για το θέμα αυτό της διατήρησης του Σολομού στα πλαίσια του πολιετούς προγράμματος, πολιετούς σχεδίου για το απόθεμα Σολομού ως και ο έχω ήδη κάνει κάποιες ε, παρατηρήσεις μέσω των τροπολογιών και θα ήθελα να πω και τα εξή. Οι 6, 7 και 13 αλλά και 17 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, διότι το όλο οικοδόμημα της τεχνικής αλίας θα πρέπει να καλυφθεί Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχολιάζει μόνο εν μέρη το θέμα της ερασιτεχνικής αλίας. Επίσης το 25, το άρθρο 25, μπορεί να είναι μια πολύ καλή ένδειξη για την κατάσταση ενός αποθέματος. Όταν υπάρχει ένας και μόνο δείκτης όμως, <clears throat> θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι λείπει κάτι, χρειάζεται ένα συμπλήρωμα. η επιστροφή των ε, Σολομών λόγω χάρη στο σημείο αφετηρίας ε, στα ποτάμια είναι κάτι σημαντικό. Τα θηλυκά επιστρέφουν, αυτό θα μπορούσε να είναι ένας Τώρα για το 18 και το 19. Και εδώ θέλουμε να δούμε κατά πόσο μπορούν να προβληθούν ηλεκτρονικά νεολόγια για όλα τα σκάφη. Ο εισηγητή δεν θέλει να είναι υποχρεωτική αυτή η καταγραφή των σκαφών, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν και διοικητικά άχθη. Τελευταίο σημείο Σε σχέση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα πρέπει να μας πούν τελικά τι θέλουν να κάνουμε με την αλία του Σολομού. Α, ε, θα έχουμε πάυση της εμπορικής αλίας Σολομού στο μέλλον. Διότι συμφωνώ ότι δεν είναι όλη η αλία Σολομού δηλωμένοι, αλλά δεν πρέπει να πλήξουμε για αυτό το λόγο και τους ε, αλείς που έχουν δηλωθεί. Καλύτερος έλεγχος της αδήλωτης αλίας. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε καλύτερα την επιβίωση του είδους. Ευχαριστούμε κύριε Κρίστερσεν, κύριε Λαβίν. Thank you, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Γκρόμπατσικ, για το έργο του. Ξέρω ότι εργάστηκε σκληρά. Εγώ τίνω να συμφωνήσω με τη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Μιλάμε για μια έκθεση και ένα πολιετές σχέδιο που σκόπο έχει να οδηγήσει στην αποκατάσταση των ε, άγριων ε, αποθεμάτων της Βαλτικής, όπως τη Σουηδία. Που έχουμε πολλά ποτάμια πλούσια σε σολομούς. Πρέπει να αποκατασταθούν λοιπόν ε, τα ποτάμια αυτά στη ροή τους, ώστε να μπορεί και ο σολομός να ανέλθει προς τις πηγές. Εδώ λοιπόν η αποκατάσταση των ε, αποθεματών είναι ο μόνος τρόπος να αποκαταστήσουμε τον άγρο σολομό. Το 70% του σολομού είναι σολομός αποκατάστασης. Και ε, ο στόχος δεν είναι μόνο να βοηθήσουμε και να εξυπηρετήσουμε την ε, βιομηχανία της αλίας, αλλά να αποκαταστήσουμε, να προστατεύσουμε τον άγριο σολομό. Διότι οι αλίες δεν γνωρίζουν αν είναι ο σολομός που ψαρεύουν άγριος ή προϊόν αποκατάστασης. Όσο για τον κύριο Βαουέσα, να και τα σχόλιά του, να πω ότι και εγώ καλωσορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά θα ήθελα να μην απομακρυνθούμε πολύ από την πρόταση της Επιτροπής, ιδίω για την αποκατάσταση και τη σταδιακή πάυση της σε 7 χρόνια. Εδώ θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο ότι η αποκατάσταση Πρέπει να γίνεται με βιολογικά αποθέματα από τον ίδιο ποταμό ή τουλάχιστον από απόσταση ελάχιστη, όσο το δυνατόν μικρότερη. Επίση, στην έκθεσή σα γίνεται η εξή παρατήρηση. Ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν με λόγια καταστρώματα ή πρότερες ή προαναγγελίε για αυτέ τι περιπτώσει. Οι περισσότεροι αλλοί Σολομού εάν θυμάμαι καλά, στην Βαλτική θάλασσα, αλλιεύουν με πολύ μικρά σκάφη. Άρα αποκλείονται πολλοί επαγγελματίε αλλιώ από αυτέ τι απαιτήσει. Ταυτόχρονα, και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σα, προτείνεται ο καθένα να συμπεριλαμβάνεται στην προαναγγελία, στο σχέδιο και στο σύστημα ελέγχου. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό. Όπω προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλοι, όλα δηλαδή τα σκάφη θα πρέπει να έχουν λόγια καταστρώματο και υποχρέωση παραγγελία. Συμφωνώ μαζί σα ότι οι εραστέχνε αλληλεί θα πρέπει επίση να υπόκεινται σε αυτέ τι υποχρεώσει υποβολή έκθεση που τον ένα τον άλλο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να επιληθεί σε επίπεδο κράτου μέλου. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ποιο μέρο των αλλιευμάτων αλλιεύεται από ε, στέχνε ψαράδε στην Βαλτική. Προτείνεται την αναθεώρηση για την απαγόρευση των σειρώμενων δικτυών. Εδώ όμως θα έχουμε δραματική μείωση εξαιτία του σχεδίου και δεν βλέπω να το επιθυμείτε αυτό γιατί δεν άλλαξε η παράγραφος αυτή της πρότασή σας. Θέλουμε πλήρη απαγόρευση των αλλιευμάτων στην ανοιχτή θάλασσα. Διότι ο μόνος τρόπος να πάνε τα ψάρια πίσω στα αποθέματα για να αποκατασταθεί και το συνολικό απόθεμα είναι να πάνε προς, τις, ε, προς το στόμα των ποταμών η Σολομή. Άρα δεν γίνεται να υπάρξουν παρασυρώμενα δίχτυα στα στόμια των, στις εκβολές των ποταμών. Αυτό είναι τελείως απίθανο. Να τη δούμε λοιπόν αυτή την απαγόρευση. Ε, η απαγόρευση που δεν ε, εισήχθη για να σώσουμε το Σολομό, αλλά αλλά για ένα άλλο είδος της Βαλτικής. Σε ό,τι αφορά τις φώκες και τους κορμοράνους, γνωρίζουμε ότι η Ελία στην ανοιχτή θάλασσα είναι ιδιαίτερα καταστρεπτική για τον αγροσολομό. Ήδη η σταδιακή μείωση θα προσφέρει πολύ περισσότερα για τη, κατά της νησιμότητας και υπέρ των αποθεμάτων σολομού παρά να δούμε τι θνησιμότητα προκαλούν οι φώκες και οι κορμοράνοι που τρώνε τους σολομούς. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό λοιπόν στο πολιτέ σχέδιο διαχείρισης να προβλέψουμε κάτι τέτοιο. Και κάτι ακόμα, που το ενέκρινε και η Επιτροπή ΕΝΒΗ και το βρίσκω άκρος σημαντικό είναι η εναρμόνιση του μεγέθους ε, εκφόρτωσης για την θαλάσσια πέστροφα και τον Σολομό. Διότι στη Βαλτική το Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Βαλτικής απίφθινε επιστολή λέγοντας ότι υπάρχουν ε, υποψίες για ε, εσφαλμένη υποβολή εκθέσεων και για το μέγεθος το, τόσο της Πέστροφας όσο και του Σολομού. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα παραθυράκι επικίνδυνο. Πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση του ελάχιστου μεγέθους ε, εκπορτωσής και για τη θαλάσσια Πέστροφα και για το Σολομό, ώστε να προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Διότι αλλιώς θα μπερδευτούν πολύ τα πράγματα. Επίσης αναφέρεστε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Βαλτική. Λέτε ότι δεν στηρίζει το σχέδιο. Εγώ προσπάθησα κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση να βρω έγγραφα από τον ιστότοπο του ΡΑΚ, του Περιφερειακού Συμβουλίου της Βαλτική. Δεν το βρήκα όμως πουθενά αυτό, να λένε ότι δεν στηρίζουν το πολιτέ σχέδιο. σα ίσα το μόνο που λένε είναι ότι δεν μπόρεσαν ακριβώ να το αποτιμήσουν ε, παρκώ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έκανε κάποιε δηλώσει για τη μερολόγια καταστρώματο, αλλά καθόλου για την προαναγγελία. Θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσετε, εάν γίνεται από αυτού. Νομίζω, λίγο πολύ, αυτά είχα να πω. Ναι. Να σας ρωτήσω και αν δέχεστε παράταση της προθεσμίας είναι πολύ αυστηρή μέχρι τη Δευτέρα. Δεν νομίζω να προλάβουμε τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λαβέν. Ο κύριος Κούν. Ορισμένες παρατηρήσεις επιπλέον για την παρουσίαση του κυρίου Γκρομπάρτσικ και του συναδέλφου Βαλέσα. Οι παρουσιάσεις αυτές πραγματικά έχουν ασχοληθεί με τα σημαντικά θέματα, με τον πληθυσμό του Σολομού και το πώς μπορούμε να τον επαναφέρουμε σε λογικά επίπεδα. Να πω ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη ε, ψαριά εξακολουθεί να μετριέται σε τόνους. Και πρέπει να δούμε πρώτα σε τι κατάσταση βρίσκεται ο πληθυσμός του Σολομού, εκεί όπου ψαρεύεται. Και φυσικά ξέρετε ότι οι καλύτερες ψαριές ε, πραγματοποιούνται εκεί πέρα όπου αναπαράγονται τα ζώα αυτά. Και αυτό το ξέρουν και οι ερασιτέχνες ψαράδες και οι επαγγελματίες ψαράδες. Και τώρα η αλία, η ερασιτεχνική αλία χρειάζεται έναν σαφέστερο ορισμό. Τι θεωρούμε ερασιτεχνική αλία, αλία αναψυχής κύριος, εάν ακολουθήσουμε την άποψη του κυρίου Γκρομπάρτσικ, τότε θα έχουμε ενδεχομένω προβλήματα στον έλεγχο. Τώρα, ο άγριος Σολωμός, η αναπαραγωγή, για, να μπορεί να αναπαραχθεί ο άγριος Σολωμός, οι συνθήκες είναι πολύ πολύπλοκες. Πρέπει να προσέξουμε πολλά επιμέρους σημεία, να δούμε πώς θα επανισάγουμε τον άγριο Σολωμό στα ποτάμια αναπαραγωγής του για να μπορέσει να ανακάμψει. Εκεί όπου παρατηρούνται μεγάλες συγκεντρώσεις ε, ψαριών, δεν ξέρουμε, μόνο τι, δεν ξέρουμε μόνο εμείς ότι είναι καλύτερο να τα λιεύσουμε εκεί, εδώ ξέρουν και οι φώκες. Μπορείτε να ρωτήσετε και να δείτε οποιαδήποτε επιστημονική μελέτη, όπως είπε η κυρία Λόβιν, ε, αυτό το απέδειξε και το Ινστιτούτο βαλτική στο Ροστόκ αλλά και στο Κίελο όπου παρατηρούνται σε αυτές τις περιοχές μεγάλες συγκεντρώσεις φωκιών. Και για ποιο λόγο. Και πότε μαζεύονται αυτές οι φώκες όταν ο Σολεμός είναι έτοιμος να ανέβει στα ποτάμια. Τότε οι φώκες πραγματικά στείλουν καρτέρι σε αυτές τις περιοχές, στα δέλτα του ποταμού και περιμένουν. Και μια χαρά ψαριά κάνουν οι φώκες. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με τον πληθυσμό της φώκιας και του κορμοράνου και πώς θα τους φέρουμε σε συνετά επίπεδα. Ε, παλαιότερα τις πυροβολούσαν. Ε, τώρα αυτό με το ημερολόγιο καταστρώματος ακούγεται μια χαρά, ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα 15 μέτρα είναι προϋπόθεση για να υπάρχει μερολόγιο καταστρώματος. Φανταστείτε τώρα, έχετε ένα πιο μικρό καίκι, τι γίνεται εκεί. Τα σκάφη μέχρι τα 12 μέτρα θεωρούνται μικρής κλίμακας αλία. Χρειαζόμαστε γι' αυτό λοιπόν ακόμα περισσότερα σχέδια διαχείρισης και για το γάδο και για το σολομό και φυσικά καλύτερη εφαρμογή τους. Και καλύτερη μετάδοση πληροφοριών. Έτσι ώστε να Και χρειαζόμαστε και καλύτερο έλεγχο έτσι ώστε οι ψαρόβαρκες να μπορούν να μεταδίδουν κατευθείαν τις πληροφορίες τους από εκεί που βρίσκονται στα διάφορα λιμάνια πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Όλα τα σκάφη, λέτε, πρέπει να έχουν ημερολόγιο καταστρώματος. Τι, και τα σκάφη που ειναι τρία, τέσσερα μέτρα, οι ψαρόβαρκες. Εκεί πέρα όπου ο ψαράς είναι πνιγμένος με ψάρια μέχρι το λαιμό, πρέπει να, έχει, να τηρεί ημερολόγιο καταστρώματος. Άλλο 12 μέτρα και άλλο μικρή βαρκούλα. Αυτά. Αλλά Τη διάθεση μου την μετέφερε η συνάδελφο εδώ δίπλα μου. Βέβαια όλα τα καλά, όλα τα κακά η κυρία Φράγκα εδώ πέρα. Ό,τι στραβό συμβαίνει εδώ η κυρία Φράγκα φταίει. Εν πάση Για την τροπολογία 25 θα ήθελα να πω κάτι και για τα σειρώμενα πλάδια. Είμαι κατηγορηματικά κατά της τροπολογίας, γιατί ήδη τα σειρώμενα δίκτυα έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Και σε καμία περίπτωση μετά από τα δεινά που περάσαμε για το θέμα αυτό να, να ξανανοίξουμε αυτό το ζήτημα. Είναι σαν να ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας. Είμαι ριζικά κατά της τροπολογίας 25 του κ. Γκρομπάρτσικ δεν ζητάει άλλο κανεί το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν το επιθυμεί. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η σειρά μου τώρα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε και για την έκθεση που στα κυριότερα τη σημεία υποστηρίζει την πρόταση της Κομισιόν για να διασφαλιστεί η συντήρηση του αποθέματος Σολομού. Ορισμένες τροπολογίες υποστηρίζουν την πρόταση της Κομισιόν για την συντήρηση των αποθεμάτων Σολομού, για παράδειγμα, οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, οι ψαριές που πρέπει να συμπεριληφθούν στις ποσοστώσεις. Όλα αυτά συμφωνούν με, την, ε, για τη, με τη συντήρηση των αποθεμάτων. Δεν θα ασχοληθώ λοιπόν με αυτές, αλλά υπάρχουν κάποια άλλα σημεία με τα οποία έχουμε κάποιες δυσκολίες. Και θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία αυτή για να σας εξηγήσω τη λογική μας πίσω από αυτή την πρόταση. Αρχίζω με τον κανονισμό για το σημείο, για παράδειγμα, που αφορά τα ημερολόγια καταστρώματος και τις ειδοποιήσεις, που είναι κάτι που, είναι αρκετά αντιφατικό, όπως είδαμε εδώ. Το σχέδιο διαχείρισης μα σκοπεύει να καλύψει όλες τις περιοχές και να συντάξει μια υπηρεσία, μια αρχή επιθεώρησης για τον Σολομό. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σολομού αλλιεύεται από μικρά σκάφη και αυτή τη στιγμή τα μικρά αυτά σκάφη δεν ελέγχονται, δεν παρακολουθούνται. Υπάρχουν τεράστια ποσοστά σολομού που αλλιεύονται κάθε χρόνο. Ένα από τα σημεία που, αναφέρει, που ανέφερε η Επιστημονική Επιτροπή στη συμβουλή, ε, στο συμβουλευτικό έγγραφο είναι η έλλειψη δεδομένων και η έλλειψη ελέγχου που οδηγούν σε προβλήματα στη διαχείριση των αποθεμάτων. Εάν δεν τα λάβουμε υπόψη, θα έχουμε χάσει ένα ποσοστό γύρω στο 9% των σκαφών που αλλιεύουν στο λαιμό. Και γι' αυτόν τον ε, λόγο αναφερθήκαμε στο στην ε, ύπαρξη ημερολογίου καταστρώματος για σκάφη πάνω από 10 μέτρα, για να καλύψουμε ακόμα περισσότερα σκάφη. Ίσως η πρότασή μας ήταν πολύ ριζική, αλλά πραγματικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα εδώ και να αναγνωρίσουμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της Βαλτικής θάλασσας είναι αυτά τα πολύ μικρά σκάφη και πολλά από αυτά τα μικρά σκάφη που ενεργοποιούνται στην περιοχή. Επίσης, με την πρότασή μας, καλύπτουμε τα σκάφη που είναι πάνω από 8 μέτρα. Ας το σκεφτούμε, λοιπόν. Η κύρια πρότασή μας ήταν η προσπάθεια να επιτύχουμε βιώσιμα αποθέματα σολομού και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε περισσότερες στατιστικές περισσότερα στατιστικά στοιχεία για να δούμε τι γίνεται, για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις. Αν όμως δεν ξέρουμε τι γίνεται, επειδή έχουμε αποκλείσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των σκαφών που θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε, θα είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Γι' αυτό και αναφέραμε το ημερολόγιο καταστρώματος. Ένα από τα άλλα ζητήματα είναι το docking, είναι η προσάραξη. Ο δεύτερος κύριος στόχος τώρα της πρότασής μας είναι να διατηρηθεί η γενετική βιοπικιλότητα του άγριου Σολομού και για να γίνει αυτό χρειάζεται σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες, να σταματήσουμε την αναπλήρωση των αποθεμάτων στα ποτάμια. Μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρόταση του εισηγητή όταν είπε ότι χρειάζονται 10 χρόνια σταδιακής μείωσης μέχρι να φτάσουμε στην απαλυφή αυτής της πρακτικής. Θα είναι δύσκολο όμως να τη συνδέσουμε με την επίτευξη του στόχου. Είναι ένας αρκετά φιλόδοξος ε, στόχος αυτός που προτείνει ο εισηγητής και για να γίνει αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τον επανεμπλουτισμό των αποθεμάτων Σολομού. Αλλά αυτό δεν μπορεί να διατηρήσει την ε, γενετική βιοποικιλότητα των αποθεμάτων. Μετά, αφορά τους ελέγχους εκφορτώσεων και το 50%. Το, το ισχύον ποσοστό επιθεώρησης είναι διαφορετικό με αυτό που προτείνουμε. Αυτό που προτείνουμε όμως, η αύξησή του, ε, αυτό που προτείνετε μάλλον εσείς, θα δημιουργήσει επιπλέον σημαντικό διοικητικό φόρτο. Κάτι άλλο τώρα. Στον ορισμό της ε, ερασιτεχνικής αλίας Τη αλίας αναψυχής. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να δώσουμε έναν λεπτομερέστερο ορισμό, αλλά εδώ θα σας προτείνω να αναφερθούμε στον ορισμό που υπάρχει στον ε, ισχύοντα κανονισμό, έτσι ώστε να αποφύγουμε τους πολλαπλούς και διαφορετικούς ορισμούς της ερασιτεχνικής αλίας. Μετά η ανάκληση της εξουσιοδότησης στα κράτη-μέλη. Αυτό συζητιέται αρκετά στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Θα ήθελα να σχολιάσω την πρότασή σας να εφαρμοστεί το άρθρο 258. Να πω ότι αυτό το άρθρο προβλέπεται να ακολουθηθεί σε περιπτώσεις παραβίασης ευρωπαϊκών νόμων. Και ως κατά συνέπεια θα υπάρχουν κυρώσεις που θα μπορούν να επιβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτή η διαδικασία είναι αρκετά γραφειοκρατική. Το να γίνει δηλαδή ανάκληση της εξουσιοδότησης των κρατών μελών. και μετά αντιμετωπίζουμε λοιπόν πρόβλημα στην ανάκληση γιατί χρειάζεται να ασχοληθούμε με, την, με τον επανεμπλουτισμό των αποθεμάτων πολύ γρήγορα. Η διαδικασία όμως ανάκλησης είναι πολύ μακρά. Δεν θα μας ε, δώσει τη δυνατότητα να αντιδράσουμε πολύ γρήγορα όσον αφορά τον επανεμπλουτισμό. Τώρα για τους θηρευτές και για τους κορμοράνους. Ε, θα το συζητήσουμε πολύ αυτό, αλλά να πω ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν δικά τους μέτρα για να ελέγξουν τον πληθυσμό των κορμοράνων. Σύμφωνα πάντα με την οδηγία για τα πουλιά. Πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα για τις επιπτώσεις που έχουν οι κορμοράνοι στο Σολομό και οι άλλοι θηρευτές στο Σολομό. Αλλά να πω ότι η έρευνα που έγινε πέρυσι δεν είχε καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα. Χρειάζεται περισσότερες μελέτες και είναι πολύ δύσκολο να αναλάβουμε δράση χωρίς ξεκάθαρα αποτελέσματα από τις μελέτες αυτές. Γι' αυτό λοιπόν θα με τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράσεις οι οποίες όμως θα επιτρέπονται και θα είναι σύμφωνες με την οδηγία για τα πουλιά. Τέλος, για την απαγόρευση των σειρώμενων διχτυών. Η απαγόρευση αυτή συνδέεται με το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ζήτησε και αυτή την απαγόρευση είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει τη δέσμευσή της ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών. Και πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε την συμμόρφωση με αυτό το ψήφισμα και να συνεχιστεί η απαγόρευση των σειρώμενων δικτυών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εν κατακλείδη να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γκρουμπάρτσικ για να τελειώνουμε και τη συζήτηση. Προτάθηκε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή τροπολογιών. Αν συμφωνεί και ο εισηγητής μας, αντί να λίγη στις 4 ε, Ιουνίου η προθεσμία για τις τροπολογίες, να την ε, παρατείνουμε μέχρι τις 11 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Οπότε αντί να ψηφίσουμε στις 20 στην Επιτροπή, θα ψηφίσουμε 11 και 12 Ιουλίου στην Επιτροπή, αφού α, ε, μας παίρνει. Εντάξει, παρατείνουμε λοιπόν την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 11 Ιουνίου 12 το μεσημέρι. Κύριε Σιγητά, ελπίζω να συμφωνείτε και έχετε το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια όλους τους συναδέλφους ε, που υπέβαλαν παρατηρήσεις και σχόλια για την έκθεσή μου. Δυστυχώς σε ορισμένα σημεία θα χρειαστεί να διαφωνήσω. Ε, μάλιστα για θέματα που είναι προφανή με βάση τη λογική που ακολουθούμε. Το πρώτο θέμα είναι η γνωμοδότηση του ΡΑΚ, του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Εγώ δεν ήμουν προσωπικά στη συνεδρίαση του ΡΑΚ, αλλά ήταν ε, προσωπικά ο συνεργάτης μου εκεί και τα άκουσε όλα. Οπότε μου λέτε ότι κάτι, ήταν διαφορετική γνωμοδότηση του ΡΑΚ, τότε τι να σας πω, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, ο συνεργάτη μου ήταν παρόν στη σύσκεψη του ΡΑΚ, του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, και ξέρω ποιο είναι το περιεχόμενο τη γνωμοδότηση και διαφέρει ριζικά από τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, το θέμα της κατάργησης ε, ε, του επανεπλουτισμού και το θέμα της ε, βιοπικιλότητας και τη ε, προστασία τη γενετικής ε, κληρονομιάς. Τώρα, αν το θέμα του επαναπλατισμού στην Βαλτική και στη βορεια θαλασσα Θάλασσα κρατάει 20-25 χρόνια, πού είναι αυτή η αγρισολομή, μια και 25 χρόνια πριν, 20 χρόνια ε, πριν είχαμε τον επανεμπλουτισμό, φτάσαμε στο, στο επίπεδο παραγωγής και τώρα μιλούμε για τεχνική αναπαραγωγή. Μα θέλουμε να διασφαλίσουμε τους άγριους ολομούς και ακριβώς ε, με την παράταση του επανεμπλατισμού είχαμε την ανασύσταση των ε, πληθυσμών των άγριων σολομών. Ούτε μπορούμε να επιτρέψουμε να υπερισχύσει ε, να δεσπόζει παντού ο νορβηγικός Σολομός. Και αυτό θα συμβεί αν μειώσουμε τους πληθυσμούς του Σολομού, που ούτως ή άλλως σε αυτό θα γεννηθούμε. Και τα σειρώμενα απλάδια του Σολομού, για, για την αλία Σολομού, αν δεν κάνω λάθος, ε, ε, εισήχθηκαν το 2008. Το 2007 είχαμε το ψήφισμα. Και έκτοτε δεν χρησιμοποιούνται σειρώμενα γελία σολομού στην Βαλτική. Και παρόλα αυτά μειώνονται ε, τα κοπάδια σολομού. Άρα δεν μπορείτε να μας λέτε ότι τα σειρώμενα απλά διευθύνονται για τη μείωση των αποθεμάτων σολομού. Ε, η κατάργηση των ε, παρασυρώμενων δικτυών θεσπίστηκε για την προστασία των δελφινιών. Ε, άλλωστε τα σειρώμενα του Σολομού ε, ε, ρίχνονται στην ανοιχτή θάλασσα. Δεν επηρεάζουν καθόλου, ούτε υπάρχει κίνδυνο να εμπλακούν στα δίχτυα αυτά η μαρσουίνη, ένα είδο φώκια. Μην μου λέτε λοιπόν ότι η απαγόρευσή του θα σώσει τα κοπάδια δελφινιών και μαρσουίνων. Ούτω ή άλλω τα πλάτια που χρησιμοποιούνται, τα παρασυρώμενα για του σολομού, δεν δημιουργούν κανένα κίνδυνο για του μαρσουίνου. Οπότε αυτό το σημείο, το σημείο της ε, επαναφοράς της χρήσης ε, των σειρώμενων απλαδιών ούτε θα εξαλείψει τον πληθυσμό Σολομού, ούτε θα απειλήσει τον πληθυσμό Μορσουίνων. Θα ήθελα παρακαλώ αυτές ε, οι αντικειμενικές ε, επιστημονικές πληροφορίες να ληφθούν υπόψη. Γι' αυτό και υπέβαλα τη σχετική τροπολογία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο. Παρακαλώ, σκεφτείτε το. Κάποιος έχει ε, και, λέμβο με κινητήρα ή έχει μια μικρή τράτα και ενώ έχει μια μικρή λέμβα με κινητήρα, τον υποχρεώνουμε να κρατάει ημερολόγιο πλοίου. Εγώ είμαι υπέρ του ελέγχου και της αεραστεχνικής αλίας, αλλά επαναλαμβάνω σας παραπέμπω στην έκθεση της, του Οργανισμού Ελέγχου της Αλίας του Βίγκο, για να δείτε πώς γίνονται οι έλεγχοι στην Βαλτική. Μερικές, μερικά σκάφη ελέγχονται τακτικά, μερικές φορές και 90%, 90 των εκφορτώσεων ελέγχονται, ενώ οι μικρές ψαρόβαρκες δεν υπάρχουν σε κανένα έλεγχο. Κάποιες λέμβοι διαφεύγουν τελείως του ελέγχου. Εγώ προτείνω 50% των εκφορτώσεων όλων των ε, λευτικών σκαφών να ελέγχεται. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, για να βελτιώσουμε τον έλεγχο. και να διαφυλάξουμε τα θέματα του Σολομού. Νομίζω ότι έτσι θα εξασφαλίσουμε τη ρίση του νόμου, γιατί όλοι έχουν υποχρέωση ε, δήλωση των αλλιευμάτων τους. Γιατί να το περιορίζουμε μόνο στους επαγγελματίες αλλιείς. Θα πρέπει να το επεκτείνουμε και στους ε, ερασιτέχνες αλλιείς. Αλλά να μην απαιτούμε από τον κάθε τουρίστα που θέλει με το καλάμι του να αλλιεύσει υποχρεώνουμε κρατάει ημερολόγιο πλοίου θα πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία εδώ και μια αναλογία. Τώρα το θέμα των θηρευτών, των φυσικών εχθρών των αποθεμάτων Σόλωμου. Εδώ το πρόβλημα είναι ακόμη πιο σοβαρό, πιο δύσκολο και πιο επίμαχο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μετακυλήσει την ευθύνη στα κράτη-μέλη. Και αυτό φαίνεται λογικό, γιατί φυσικά κανένας δεν θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη για το τόσο επίμαχο θέμα. Και την ε, επιρρύπτει σε άλλον. Αλλά από γεωγραφική άποψη είναι δύσκολο τα κρατημέλη από μόνα τους ε, να εφαρμόσουν διάφορα σχέδια διαχείρισης. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, συνεχίζεται η διαδικασία της ανασύστασης με βάση τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανασύστασης ε, του αποθέματος γκρίζα φώκιας. Ενώ στην Σουηδία, δεν κάνω λάθος, στη Φιλανδία, όπως ακούσαμε χθε και από σας το άκουσα, ε, έχει, είναι πολύ μεγαλύτερα. Η γκρίζα φώκια στην ε, Σουηδία-Φιλανδία είναι πολύ πιο παρούσα και, και πραγματικά έχει ολέθρια συνέπεια για τα αποθέματα Σολομού. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε ότι το θέμα της αντιμετώπισης θηρευτών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε κράτους. Είναι αδύνατο το κράτος μέλος από μόνο του να τα βγάλει πέρα. Γι' αυτό και διαφωνώ με την σχετική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά. Αυτά προς το παρόν. Θα έχω φυσικά και προσωπικές συνομιλίες. Θα συνεννοηθώ με τους συναδέλφους και σας παροτρύνω να καταθέσετε τις τροπολογίες σας για να εμπλουτιστεί η έκθεση. Ωραία. Περνούμε στο 22. Διάφορα. Δεν υπάρχουν. 23. Ανακοινώσει του Προέδρου ως προς τις αποφάσεις των συντονιστών. Έχω μεταβιβαστεί ήδη. Αν δεν υπάρξουν αντιρρήσει, θα θεωρηθούν συγκεκριμένε οι αποφάσεις των συντονιστών. Η επόμενη μα συνεδρίαση θα γίνει 20 Ιουνίου πρωί και απόγευμα και 21 Ιουνίου το πρωί μόνο. Αυτά, σα ευχαριστώ. Εξαντλήσαμε τα σημεία τη ημερήσια διάταξη. Ήταν πολύ έντονο αυτό το διήμερο. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, τη γραμματεία, τους διερμηνείς και το καθεξής και ραντεβού στην επόμενη μας συνέδρια Υπότιτλοι